Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Με κάποια καθυστέρηση μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ο συνήθως, τις Δευτέρες. Είναι η μέρα που έρχονται οι ευρωβουλευτές από τις χώρες τους. και γι' αυτό καθυστερούμε και συνήθως κρατάμε μια καθυστέρηση κατά την έναρξη της συνεδρίασης μας τη Δευτέρα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους παρόντες ευρωβουλευτές, τους καλεσμένους μας και τους ειδικού μας καλεσμένους, τους εμπειρογνώμονές μας. Αλλά πρώτα να δούμε κάποια διαδικαστικά και να εγκρίνουμε πρώτα απ' όλα την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Και έχουμε καλεσμένους του κυρίου δες Ε, ναι, δημοσιογράφη η καλεσμένη του κυρίου Ντες και θα κάνω και κάποιες μαγνητοσκοπήσεις ε, κάποιων τμήματων της συνεδρίασης. Επίσης έχουμε και δημοσιογράφους από τη Γαλλία. Από το κανάλι France 3, το γαλλικό. Θα ήθελα να καλωσορίσω και, τα δύο, και τους δύο ομάδες δημοσιογράφων. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Είναι ενδιαφέροντα τα θέματα που θα εξετάσουμε σήμερα και γι' αυτό προτείνω να περάσουμε κατευθείαν σε αυτά. Το πρώτο θέμα της απογευματινής μας συνεδρίασης είναι οι επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας στην τροφική αλυσίδα και στην κοινή γεωργική πολιτική. Πρόκειται για μια μελέτη που εκπώνησε η κυρία Μόνικα Πέσ η Μαρία Κύροβα από την ε, εταιρεία Βαλντάνη Βικάρη και Ασοσιάτη της Ιταλίας και η κυρία Κατερίν Σόμε από το ερευνητικό κέντρο Wageningen της Ολλανδίας. Το πανεπιστήμιο αυτό πολύ συχνά μας ε, εκπονεί μελέτες. Επίσης, Πρόκειται για μια μελέτη που ανατέθηκε ε, από το Τμήμα Πολιτικής Β στους εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση της μελέτης με θέμα της επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας στην τροφική αλυσίδα και την ΚΑΠ. Μάλιστα, εγκύψαμε για πρώτη φορά στο πρόβλημα αυτό το Νοέμβριο του 2017. Τότε η Επιτροπή μας ζήτησε την κατάρτιση μιας μελέτης ε, γιατί είχαμε ραγδαίες εξέλιξεις στην ψηφιακή οικονομία που επηρεάζουν ιδιαίτερος και τον κόσμο της παραγωγής, διανομής, αγοράς και πώλησης των καταναλωτικών αγαθών και των τροφίμων. Ε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 4.0 που εξελίσσεται ε, με αστρονομική ταχύτητα και επηρεάζει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας και τη γεωργία. Ε, εν ώψη λοιπόν μιας ε, βιώσιμης γεωργίας και συστημάτων παραγωγής που θα, είναι αποδο... θα κάνουν αποδοτική χρήση και αποτελεσματική χρήση των πόρων, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που δίνει η ψηφιακή οικονομία από όλη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων. Επίσης έχουμε πολύ διαφορετικές ανατρεπτικές ρηξικέλητες τεχνολογίες που επιτρέπουν ε, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ε, αλυσίδας, της τροφικής αλυσίδας. Έχουμε την ε, γεωργία ακριβία, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την αυτοματοποίηση της γεωργίας και την καινοτομία στη μεταποίηση των τροφίμων και το λιανεμπόριο. Γι' αυτό θα είναι χρήσιμε πληροφορίε και οι κατευθυντήρες γραμμές που θα λάβουμε για το δυναμικό της ψηφιακή καινοτομία, προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα την κοινή πολιτική. Όπω είπε η μελέτη αυτή ανατέθηκε και τη διαχείριση της εξασφάλισης του τμήμα πολιτικής Β. Ε, σας είπα ποιοι φορείς εκπώνησαν τη σχετική μελέτη και μάλιστα καλώς όρισα και τους εκπροσώπους, τις εκπροσώπους αυτών των φορέων. Και θα δώσω τώρα το λόγο στις εμπεργόμενες που κατάρτισαν τη μελέτη. Μεταξύ σας θα αποφασίσετε πώς θα μοιραστείτε το 20 λεπτό που έχετε για την παρουσίαση. Βέβαια, ίσως δεν είναι πολύ ο χρόνος για να μας παρουσιάσετε τόσο πολύ τη μελέτη, αλλά τίποτα δεν είναι ανέφικτο, γι' αυτό σας παρακαλούμε να είστε σχετικά συνοπτικές. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τη μελέτη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνοψίσουμε αυτή την πολύ πυκνή μελέτη που έχετε φαντάζομαι δει ήδη στην ε, πολυσέλιδη μελέτη μας, μέσα σε μερικές μονοδιαφάνειες. Ξεκινώ λοιπόν με τις κύριες στάσεις στην ψηφιακή οικονομία, τα ωφέλη και τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης, τις απόψεις των εμπλικωμένων παραγόντων, τις διάφορες πλευρές, τις ε, ανατρεπτικές τεχνολογίες που έχουμε λάβει υπόψη μέσα στη μελέτη μας, κάποιες ε, συγκεκριμένες υποθέσεις και πρακτικά, πρακτικές εκτιμήσεις, πρακτικές μελέτες, ε, τις συνέπειες στην κατακόρυφη ολοκλήρωση, τις συνέπειες στην την πολιτική και τα συμπεράσματα. Ξεκινώ λοιπόν με τις ε, κύριες τάσεις. Η ζήτηση για τεχνολογία στη γεωργία ε, αυξάνεται και μπορεί να προσφέρει δυνατότητες για το γεωργό στην αντιμετώπιση των τωρινών αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων, όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση της αγοραστικής ε, δύναμης, της ζήτησης, που σημαίνει όμως ταυτόχρονα και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και ε, αλλαγές στα μοντέλα της ε, κατανάλωσης, ζήτηση μεγαλύτερη για ε, βιολογικά προϊόντα, για ενημέρωση πληροφορίες, δηλαδή ανιχνευσιμότητα για την προέλευση των προϊόντων, για ζητήματα δυσανεξίας συστατικών. Όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η κατανάλωση καθοδηγεί την ζήτηση σε, νέες μορφές, σε νέους τύπους προϊόντων και αυτά όλα βέβαια πάντα με δεδομένες τις ανάγκες για προσαρμογή και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, το κόστος και την ανάγκη για βελτίωση παραγωγικότητας χωρίς σημαντική επιβάρυνση σε όρους κόστους. Όλες αυτές οι τάσεις λοιπόν οδηγούν σε μεγαλύτερη, σε ανάγκη για μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία. Όπως είπα, ζήτηση, απέτηση για νέα και βιολογικά προϊόντα, για ενημέρωση ο πολίτης θέλει να ξέρει από πού προέρχονται τα προϊόντα του, πώς έχουν παραχθεί, τάσεις διατροφικές, τις ε, οποίες ε, ορίζει ο καταναλωτής μέσω της αγοράς. Και επίσης η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλλει στην μεγαλύτερη ενοποίηση όλης της ε, αλυσίδας αξίας με μεγαλύτερη ροή πληροφοριών αλλά και καλύτερες καλύτερη κυκλοφορία των προϊόντων, Ενδεχομένω δεν θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργάζονται όλοι οι παράγοντε στην ε, αλυσίδα τη ε, αξία. Οι νέε τεχνολογίε φέρνουν αλλαγέ, στους τρόπους παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, ανάλογα βέβαια και με το μέγεθο τη εκμετάλλευση, αλλά και με διαφορετική στάση έναντι της ε, καινοτομίας αυτής, πάλι ανάλογα με το μέγεθος, αλλά και με την ηλικία πλέον, όχι μόνο το μέγεθος της εκμετάλλευσης, αλλά και την ηλικία του γεωργού. Η δε βιοτεχνολογία φαίνεται πως θα προσδιορίσει το μέλλον της γεωργίας με τη δυνατότητα που δίνει να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως καιρικά φαινόμενα, όπως ε, νόση, αλλά και εγείροντας ταυτόχρονα προβληματισμούς και απειλές, κυρίως σε σχέση με τις ανησυχίες του καταναλωτή. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, λοιπόν. Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να διαβάσετε τα μικρά γράμματα στη διαφάνεια, γιατί δεν ξέρω αν από την απόσταση στην οποία κάθεστε μπορείτε να το διαβάσετε. Έχουμε λοιπόν στα αριστερά τις προκλήσεις συνοπτικά ξεκινώντας όπως είπα και νωρίτερα από το ζήτημα του μεγέθους της εκμετάλλευσης, ένα μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης στην Ευρώπη που ξέρουμε ότι απέχει πολύ από τα μεγέθη που βλέπουμε στις ΗΠΑ και που επηρεάζει πολύ συχνά την κατάσταση γιατί υπάρχει απουσία γνώσεων ή δεξιοτήτων ή ε, δυναμικού επενδύσεων και έτσι ο γεωργός θα πρέπει και να είναι ε, σίγουρος για το πόσο αποτελεσματική θα είναι η καινοτομία για να την εισαγάγει, αλλά και ε, να μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο, τη διακινδύνευση από την επένδυση. Δεν μπορεί δηλαδή να σηκώσει το βάρος ε, του κινδύνου ή την αβεβαιότητα από τις επενδύσεις, γιατί ήδη έχει πολύ ψηλό κίνδυνο να λάβει σχετιζόμενο με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες. Επίσης έχουμε μια απέτηση σχετική με την ψηφιοποίηση πρωτογενή, που δεν είναι χαρακτηριστική μόνο στη γεωργία. Χρειάζεται η ε, ευρυζωνικότητα, χρειάζεται η συνδεσιμότητα ε, παντού. Και αυτό βέβαια για τις ε, περιοχές της υπαίθρου της Ευρώπης είναι ακόμη μια μεγάλη πρόκληση. Και επίσης ένα θέμα που συζητήθηκε, ξέρουμε πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, Το ζήτημα των δεδομένων, δηλαδή η διακυβέρνηση για μια ισοδίκη κατανομή των δεδομένων. Μια από τι μεγάλε προκλήσει είναι σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα, ποιο τα διαχειρίζεται. Ε, εάν, ε, και όλο αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφώσει, θα επηρεάσει δηλαδή την ψηφιοποίηση και τις εξελίξεις της. Υπάρχουν και άλλα, άλλες πιθανές, πιθανά αρνητικές συνέπειες με απώλεια θέσεων ε, εάν μιλήσουμε για αυτοματοποίηση αλλά και μονοπωλιακές θέσεις εφόσον εισαχθούν στις αγορές μεγάλοι παράγοντες, τόσο μεγάλοι που θα επηρεάσουν ε, δυσμενώς ανταγωνιστικά τις μικρότερες μονάδες. Υπάρχουν όμως και πολλά θετικά. Υπάρχει και θετικός αντίκτυπος. Ε, σε κεφάλαια σας τον παρουσιάζουμε ξεκινώντας από τους γεωργούς τους ίδιους, με την αύξηση παραγωγής, με τον περιορισμό του κόστους αυτής της παραγωγής, με την ε, υποστήριξη αποφάσεων χάρη σε δεδομένα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί έτσι επιτρέπεται και η πρόβλεψη ακόμη και των καιρικών συνθήκων και η βελτίωση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου για τον καταναλωτή. Επίσης έχουμε δεδομένα και πληροφορίες παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Για τις δημόσιες αρχές, το τρίτο κεφάλαιο, τα ωφέλη είναι πιο ασφαλή δεδομένα για την αξιολόγηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων και αποτελεσματική λειτουργία της κοινωνικής πολιτικής. Για το περιβάλλον έχουμε τον περιορισμό της ε, κατανάλωσης ύδατος, αλλά και ε, την χρήση, καλύτερα, καλύτερη χρήση, πιο οικονομική χρήση, όχι μόνο των υδάτων, αλλά και των ε, ζυζανιοπτρών και λοιπόν στοιχείων που χρησιμοποιεί η γεωργική η οικονομία και άρα είναι καλύτερα για το περιβάλλον. Έχουμε ταυτόχρονα και τους νέους παράγοντες που εμφανίζονται στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι οι νέες επιχειρήσεις, αγροτεχνολογικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερη ε, ιδιαίτερα σημαντικέ ευκαιρίε για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις με νέες τεχνολογίες και παραγόντες που μπαίνουν στο χώρο των ε, ε, γεωργικών τροφή, της γεωργίας και των τροφίμων και την ανάπτυξη νεοφιών επιχειρήσεων. Άρα είναι πολλά και σημαντικά τα ωφέλη. Οι παράγοντες, λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι στην αλυσίδα της αξίας πολύ και ξεκινώ πρώτα από τον γεωργό και τον προμηθευτή του γεωργού για να ξεκινήσω καλύτερα. Δηλαδή εδώ έχω να κάνω με αυτόν ο οποίος έχει να αναπτύξει νέες δυνατότητες και να εισαγάγει στην, στον τρόπο εργασίας του την τεχνολογία, η ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας σημαίνει και καλύτερη συλλογική δεδομένων και βαθύτερη ανάλυση αλλά και επιμερισμό των πληροφοριών που επηρεάζει οπωσδήποτε και τον προμηθευτή του Γεωργού. Ταυτόχρονα αυτό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται αυτή η επιχείρηση προμήθειας γεωργικών προϊόντων ε, της δουλειάς της και βέβαια θα επηρέασε αντίστοιχα και τους λοιπούς παράγοντες. Για το Γεωργό. Ο Γεωργός δεν είναι πάντα δετεθειμένος να εισαγάγει ανεφετέρου την ψηφιοποίηση. Όπως είπαμε στην αρχή ε, της διαδικασίας της καινοτομίας, ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, είναι αρκετά υψηλός. Άρα θα έχουμε τον πιο καινοτόμο αυτόν δηλαδή που θα επιλέξει την καινοτομία στην αρχή και εκείνον τον Γεωργό, ο οποίος θα ακολουθήσει μόνο άπαξ και αξιολογηθεί ως αξιόπιστη η τεχνολογία αυτή και άρα θα έχει τη θεσή του αξιόπιστες πληροφορίες πως θα είναι ωφέλιμη για αυτόν η εισαγωγή της ε, καινοτομίας αυτής. Άρα η διαδικασία εισαγωγής νέας τεχνολογίας είναι αρκετά βραδία, δεν παρασύρει στην πορεία της όλους τους γεωργούς και πάντως δεν τους παρασύρει ταυτόχρονα. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργηθεί αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνης και εξοπιστίας. εμπιστοσύνης. Ε, η, η διανομή και το λιανεμπόριο που ζητεί την εισαγωγή ανιχνευτών για τη συλλογή πληροφοριών που θα αξιοποιήσουν, προσφέροντας έτσι περισσότερες πληροφορίες βέβαια στον καταναλωτή αφενός. Αφετέρου όμως και στο πλαίσιο της ε, ψηφιοποίησης μπορούμε να δούμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο με το οποίο μπαίνουν νέοι παράγοντες στην αγορά, παράγοντες που δεν δραστηριοποιούνταν στην αγορά των γεωρικών προϊόντων και άρα ως εκ τούτου και αλλάζουν την αλυσίδα αξίας αλλά και τα επιχειρηματικά μοντέλα με τα οποία, τα οποία ήταν μέχρι τώρα γνωστά και αυτό επηρεάζει βέβαια και το επιμελητιακό σκέλος για τα οποροκυπευτικά, για τα οπορολαχανικά, επιτάχυνση των διαδικασιών με λιγότερα, λιγότερα προβλήματα και άρα καλύτερη ποιότητα του προϊόντος που φτάνει στο καταναλωτή. Ο δε καταναλωτής και θα έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με το παρελθόν. Και θα χαράζει τις τάσεις με τις επιλογές του, όπως είπαμε, βιολογικά προϊόντα, τοπική παραγωγή, όλα αυτά τα οποία απαιτεί να έχει πλέον με ο καταναλωτής ε, ως πληροφορία και χάρη στην ψηφιοποίηση και αντιστοίχω επηρεάζουν τις διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Οι νεοφύης επιχειρήσεις ανεφέρθησαν και νωρίτερα, είναι οι παράγοντες ε, στην αγορά της Ευρώπης που εξαρτώνται και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε τις νεοφύης μόνο μέσα στη Monsanto, την Bayern, την BASF, δηλαδή μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ τώρα έχουμε μικρότερη επένδυση σε όγκο, αλλά απέτηση να ε, προσφέρεται η παραγωγή της καινοτομίας από τις μικρομεσαίες, από τις νεοφυείς, αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, έξω από τους γίγαντες. Άρα προτιμάω η μεγάλη επιχείρηση όχι να αναπτύσσει πλέον εσωτερικά την καινοτομία, αλλά να την εισαγάγει άπαξ και αυτή επικυρωθεί. Αυτό το βλέπουμε ήδη να εμφανίζεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Ευρώπη λιγότερο ε, εμφανές ακόμη, αλλά είναι σαφές πως έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ειδικευμένε στη γεωργία και κάποιες μικρές νεοφύσεις οι οποίες αναπτύσσουν την καινοτομία. Διεθνείς και κυβερνητικοί οργανισμοί επίσης με σαφείς στόχους θέλουν, θέλουν την ε, ψηφιοποίηση για να στηρίζουν τους γεωργούς και να αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά προβλήματα περιορισμό, δηλαδή στην ε, καταναλώση του, στη χρήση των ζανιοκτώνων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, βελτίωση ή περιορισμό των, ε, του αντικτύπου της γεωργικής παραγωγής ε, στο περιβάλλον, βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων, της προμήθειας σε τρόφιμα. Όλα αυτά μπορεί η ψηφιοποίηση να τα υποστηρίξει. Και υπάρχει βέβαια και η επιστημονική θεώρηση ο επιστήμονας που ζητεί την πρόσβασιμότητα σε όλα αυτά τα δεδομένα και έτσι θα έχει καλύτερη ε, και πρόσθετη γνώση και άρα παραγωγή και νέας καινοτομίας. Και εδώ δίνω το λόγο, αν μου επιτρέπετε, στη συνάδελφο. Ήδη στη φάση της πρότασης γίνεται διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών που έχουν ε, μεγάλο αντίκτυπο, μεσαίο αντίκτυπο ή χαμηλό αντίκτυπο. Οι τεχνολογίες με τις μεγάλες επιπτώσει περιλαμβάνουν το ίντερνετ, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την αυτοματοποίηση, η ρομποτοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την ίχνηλασιμότητα και τα μαζικά δεδομένα. Περιμένουμε αυτέ οι ανατρεπτικές τεχνολογίε ε, να επηρεάσουν ε, ιδιαίτερο στην κατάσταση και μάλιστα βράχει πρόθεσμα. Οι τεχνολογίες που μέσω πρόθεσμα θα επηρεάσουν είναι επίσης πολύ προηγμένες και θα επηρεάσουν ε, σχετικά σύντομα την κατάσταση, αλλά όχι βράχει πρόθεσμα, μέσω πρόθεσμα. Είναι κάπως αβέβαιη οι πτώση τους. Αφορούν την ε, τεχνολογία blockchain, το παγκόσμιο, σύστημα δορυφορικής, ε, το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα προήγησης, και την εικονική πραγματικότητα. Επίσης, ε, άλλα σημαντικά συστήματα που έχουν χαμηλές επιπτώσεις ε, είναι ε, ήδη καταξιωμένα, όπως η ευρυζωνικότητα, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και οι πλατφόρμες για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Έχουμε και μεμονωμένες περιπτώσεις τώρα, παρακολούθηση μεμονωμένων περιπτώσεων, που στηρίζονται σε έξυπνους γεωργικούς κόμβους, Έχουμε το 2020 που ξεκινάνε σήμερα και είναι σχετικά καινούργιες, καινούργιες τομείς μελετών και επίσης ε, βρίσκεται σε φάση πρωτόλια ακόμη. Χρησιμοποιούν ε, την κατάσταση, ε, τους αισθητήρε για την υγεία των χείρων και τη χρήση αντιβιωτικών. Επίσης τεχνητή νοημοσύνη, μαζικές, ε, μαζικά δεδομένα. Αυτές οι έρευνες γίνονται στη Γερμανία. Ένα από τα συστήματα, από τα παραδείγματα που εξετάσαμε είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνολογιών, ε, διαδίκτυο πραγμάτων, τεχνητή ε, νοημοσύνη, αυτοματοποίηση ε, και γίνεται και εντοπισμό ασθενειών, επιβλαβών οργανισμών και ιών ε, σε ελαιόδεντρα, μπέλια και φελοδρίς. Γίνεται στην Ισπανία επίσης. Ε, άλλο σημαντικό πρόγραμμα γίνεται στον μεγαλακτοκομικό κλάδο με συνδυασμό τεχνολογιών, μαζικά στοιχεία που συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, ζωοτροφές, καλλιέργειες, καιρικές συνθήκες, καλή μεταχείριση των ζώων στον γαλακτοκομικό τομέα. Και συνδυάζεται λοιπόν εδώ τα μαζικά δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, ε, η αυτοματοποίηση και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Και στην Ελλάδα είχαμε ε, συνδυασμό του ε, διαδικτύου πραγμάτων, των μαζικών δεδομένων και τις, τις τεχνολογίες τις δορυφορικές για την παρακολουθήση για παραγωγή φιλοδών λαχανικών. Επίσης είχαμε μια περίπτωση με υδροπονικές καλλιέργειες και εκεί έγιναν έρευνες διαφόρων τέτοιων σχεδίων και πέραν αυτών των τεχνολογιών υψηλού αντικτύπου έχουμε και ένα πρόγραμμα για την τεχνολογία blockchain που καλύπτει 30 προγράμματα και εκεί είχαμε χνηλασιμότητα για διάφορα προϊόντα όπως αυγά, ντομάτες, σολομό και ούτω καθεξής. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ ενδιαφέροντα για τους ε, πελάτες, ε, για τους ε, καταναλωτές και τα θέματα επίσης εικονικής πραγματικότητας είναι πολύ ενδιαφέροντα για τους καταναλωτές και άλλους φορείς αλυσίδας αξίας. Και στην περίπτωση του McDonald's του Ενωμένου Βασιλείου μπορέσαμε να δώσουμε στους καταναλωτές να δούμε τι συμβαίνει από την στιγμή της συγκομιδής της πατάτας. Επίσης, ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης, έχουμε ένα, μια χαρτογράφηση που γίνεται με drones ε, της υγρασίας του εδάφους. Επίσης, έχουμε την αλυσίδα προμηθείας για τους γεωλογικούς σπόρους και τον τρόπο βελτιστοποίηση αυτή τη αλυσίδα και σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποστήριξη, τι μεταφορέ, την αποθήκευση και τον σχεδιασμό. Ε, και την αποτελεσματικότητα φυσικά όλων αυτών των επιμέρους στοιχείων. Τι κάναμε στην ανάλυση σε ό,τι αφορά την κατακόρυφη ολοκλήρωση της αλυσίδα ε, τροφίμων είναι ότι ε, χωρίσαμε τις περιπτώσεις αυτές σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν η αποτελεσματικότητα της ε, αλυσίδα αξιών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε αποτελεσματική χρήση των ισρώων, Έχουμε την υγεία των χείρων και τις επιβλαβείς οργανισμούς για τις καλλιέργειες. Έχουμε τους χάρτες για την υγρασία του εδάφους, επίσης, που καθιστούν πιο αποτελεσματική τη γεωργία, αλλά και την περίπτωση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και την υλικοτεχνική επιρροή. Επίση, δεύτερη περίπτωση, έχουμε τι βραχύτερε αλυσίδε τη αξία. Αυτό είναι σημαντικό για τι μεγάλε εταιρείε. Εδώ περιλαμβάνουν τι υποθέσει ε, υδροπονική καλλιέργεια και τα μαζικά δεδομένα. Η τρίτη κατηγορία ουσιαστικά συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς. Και αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην τεχνολογία blockchain και την εικονική πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της κοινή γεωρικής πολιτικής, ε, κάναμε μια αξιολόγηση με βάση όλες αυτές τις υποθέσεις που εξετάσαμε, όλα αυτά τα παραδείγματα. Σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της σταθερότητας της ε, αγοράς, είναι κοινό χαρακτηριστικό, μείωση των κινδύνων και η εξασφάλιση μεγαλύτερη διαφάνεια στην ε, μετάδοση των πληροφοριών. Όλα αυτά τα στοιχεία αυξάνουν την σταθερότητα της αγοράς. Σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των προσδοκιών του καταναλωτή, και αυτός είναι στόχος της ΚΑΠ. Και με τις τεχνολογίες ε, που μειώνουν τις τιμές, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και μειώνουν τους κινδύνους, μπορούν και οι οι καταναλωτές, οι πελάτες να εξασφαλίσουν η χρησιμότητα χρησιμοποιώντας το blockchain και την η εικονική πραγματικότητα. Αλλά η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας γεωργίας και η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ήταν τα πιο θετικά ζητούμενα και στις, σε όλες αυτές τις υποθέσεις είχαμε θετική εξέλιξη. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη χρήση των ισορροών, με την μείωση της χρήσης των λιπασμάτων έχουμε θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και μία κυκλικότητα των προϊόντων, μείωση των αποβλήτων και επίσης χάρη στη χρήση της τεχνολογίας blockchain και της εικονικής πραγματικότητας εξασφαλίζεται καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Αλλά και σε ό,τι αφορά το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, και εκεί είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί με τις μεταφορές μειώνεται ο χρόνος μεταφο- στις μεταφορές μειώνεται ο χρόνος μεταφοράς, ιδιαίτερα με τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και το θέμα αυτό έχει κάποιες διασυνδέσεις και με τη χρήση των τεχνολογιών, της τεχνολογίας blockchain. Επίσης, η βιοπικιλότητα που εξασφαλίζεται με τη γεωργία και η εξασφάλιση της ανάπτυξης της υπαίθρου, γιατί αν τα αφήσουμε όλα αυτά στις αγορές μόνο, στην αυτορύθμιση των αγορών, σίγουρα δεν ε, θα υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι. και ίσως έχουμε μια αύξηση του οικολογικού αποτυπώματος στις, ε, στην Ήπεθρο. Και για να ολοκληρώσω το η τελευταία διαφάνεια με τα συμπεράσματα, ποιε είναι πιο αρνητικές αιτίε, ποιε είναι οι προκλήσεις δηλαδή που εξωθούν τους γεωργούς να στραφούν προς την τεχνολογία και την καινοτομία. Έχουμε το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τις κλιματικές ε, ε, συνθήκες που θα σε κίνδυνο τη γεωργική δραστηριότητα. Επίσης, ε, η αβεβαιότητα τη μέλλοντος της ζήτησης ε, λόγω της αστιφιλίας ε, και της απερίμωσης της υπαίθρου λόγω της αστιφιλίας. Επίσης, αύξηση του πληθυσμού και κοινωνικές αλλαγές που αναφέραμε και προηγουμένως και ανάγκη της βελτιστοποίησης παραγωγής προκειμένου να αντισταθμιστεί το υψηλό κόστος παραγωγής. Όλε αυτέ είναι αιτίε που οδηγούν ε, του γεωργού σε στι τεχνολογίε. Έχουμε και βασικέ αιτίε που επιταχύνουν ε, την προσαρμογή στην ψηφιοποίηση τη αλυσίδα αξιών. οι, ανάγκες και οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν, γίνονται πιο απαιτητικοί, ζητούν περισσότερη ενημέρωση, καλύτερε πληροφορίε. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστεί και η αλυσίδα αξιών σε αυτέ τι νέε απαιτήσει. Επίση, αναφέραμε την ευρυζανικότητα, την παρουσία καλών υποδομών, προηγμένων υποδομών που πρέπει να εφαρμοστούν. Και αυτό μπορεί να βελτιωθεί χάρη στι πολιτικέ. Επίση, προσβασιμότητα στα δεδομένα και ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα. Ποιο είναι ο κύριο των δεδομένων, ποιο τα διαχειρίζεται, ποιο τα επεξεργάζεται. Αυτό είναι θετικό παράγοντα, αλλά μπορεί να μετατραπεί και σε απειλή. Επίση, υπάρχουν αρκετέ επενδύσει στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την ε, προαγωγή τέτοιων ε, τεχνολογικών ε, εξελίξεων. Βέβαια, βρισκόμαστε ακόμη στα σπάργανα σε όλα αυτά τα θέματα και θα έχουμε πρόοδο αν έχουμε αρκετέ επενδύσει. ό,τι αφορά τι επιπτώσει στην αλυσίδα αξιών, πέραν τη ολοκλήρωση, έχουμε και άλλε επιπτώσει. Η μείωση των κινδύνων τη γεωργική παραγωγή θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία. Επίσης, οι κίνδυνοι που αφορούν και συνδέονται με τις κλιματικές απειλές, καλύτερη αποτελεσματικότητα στην παραγωγή και ανάγκη προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ε, ανάγκες των καταναλωτών, επίσης καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση νερού και ενέργειας, ενημέρωση για τις υλικοτεχνικές υποδομές σε όλη την αλυσίδα των αξιών και νέες, πιθαν... νέες δυνατότητες για τους πελάτες, για τους καταναλωτές να γνωρίζουν όχι μόνο την προέλευση των τροφίμων, αλλά και τη διαδικασία παραγωγής που οδήγησε ε, στο να έρθουν αυτά τα τρόφιμα στο πιάτο του καταναλωτή. Αυτά ελπίζω να μην μακρηγορήσαμε. Ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε τη παρουσίαση που μας κάνατε της μελέτης σας και θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Δεν είναι και πολύ εύκολο το θέμα σίγουρα. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Σάγκνη είναι ο πρώτος εγγεγραμμένος ομιλητής, αλλά συνομιλεί με τον κύριο Ταραμπέλα τώρα, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Χόισλινγκ. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχουμε ακούσει πολλά για τις νέες τεχνολογίες και τη συλλογή δεδομένων και όλα είναι υπέροχα και ωραία. Τώρα το αν έχουν όλα νόημα είναι άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον κύριο Ρος, που είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τεχνολογίας ο οποίος σε μια συνέντευξη είπε ότι οι δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών ε, υπερεκτιμούνται. Ε, με έξυπνη διαχείριση θα μπορούσε να πετύχει κανείς πολύ περισσότερα από ότι με νέες τεχνολογίες ε, και μπορώ μόνο να συμφωνήσω μαζί του. Ε, πολλές ε, ελπίδες ε, συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες. Αναφέρατε τη Monsanto, τη McDonald's, τους οποίους, τους, οι οποίοι έχουν πολλά συμφέροντα στην υπόθεση αυτή. Η Monsanto είναι μεγάλος παράγοντας, αλλά γνωρίζετε το θέμα με τις μέλισσες και όσον αφορά τα δεδομένα, ποιος θα διαχειρίζεται, πώς μπορούμε να φροντίσουμε να μην υπάρξει κατάχρηση των δεδομένων. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Δύο φορές ε, σύντομα αναφερθήκατε σε περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Ο Επίτροπος θεωρεί ότι είναι ένα από τα σημαντικά μέτρα για να ε, εξοικονομήσουμε φυτοφάρμακα. Έχετε κάποια ε, μελέτη που να το αποδεικνύει αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια. Ε, γίνονται πάντα προσπάθειες για βελτιστοποίηση των ε, τεχνολογιών ε, και των λοιπασμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μειωμένη χρήση. Μάλιστα, ο παραγωγός θέλει να χρησιμοποιήσει περισσότερα για να αυξήσει την παραγωγή του. Υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε εξοικονόμηση φυτοφαρμάκων. Εγώ νομίζω ότι αυτό ε, είναι απλά μια υπόθεση. Ε, αναφέρεται επίση η χρήση τεχνολογιών για εξοικονόμηση νερού. Υπάρχουν όμω και εδώ πρακτικέ λύσει. Δεν χρειάζεται να ε, βασιστούμε σε σύγχρονε τεχνολογίε. Υπάρχουν τεχνικέ γνωστέ εδώ και δεκαετίε. Αυτό που με ενοχλεί στην όλη συζήτηση είναι ότι η υπόσχεται πολλά η νέα τεχνολογία, αλλά πολύ συχνά τα προβλήματα που λύνουμε με την τεχνολογία είναι αυτά που δημιούργησε και η τεχνολογία. Εγώ ως ε, παραγωγός στη βιολογική γεωργία θα χαιρόμουν ε, αν οι, ε, οι γεωργοί πάνε να δούνε τι γίνεται στο, στη γη τους αντί να βασίζονται σε δεδομένα των δορυφόρων. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις ρίζες αντί να ελπίζουμε ότι η τεχνολογία θα λύσει προβλήματα τα οποία δημιούργησε και η τεχνολογία άλλωστε. Εγώ έχω αμφιβολίες εάν υπάρχουν αποδείξεις τότε εντάξει, αλλά οι ελπίδες ε, που ε, ε, εκφράζει η Κομισιόν νομίζω ότι είναι υπερβολικές. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω να μην βάλετε όλα σας τα χρήματα σε τέτοιες ε, τεχνολογίες, ε, διότι τελικά νομίζω ότι αυτοί που επωφελούνται είναι οι μεγάλες εταιρείες και όχι οι μικροί γεωργοί. Έχουμε λίγο χρόνο, οπότε έχω ένα σχόλιο. Ε, είμαι πολύ περίεργος τι θα έλεγε σε αυτά που είπατε ο κύριος Γιάν Χόιτεμα, που είναι άλλη γενιά, είναι πιο νέος και βλέπει διαφορετικά τη Γεωργία από εμάς που είμαστε κάπως πιο μεγάλοι. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες και στους νέους για να έχουν την καλύτερη, καλύτερο φάσμα επιλογών, μεγαλύτερο φάσμα επιλογών. Οπότε και τη δική του γνώμη θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Σίγουρα οι νέε τεχνολογίες είναι πολύ δαπανηρές. Και το θέμα είναι ποιο θα καλύψει αυτό το κόστος που θα αυξηθεί. Η κοινή ιερική πολιτική θα καλύψει την αύξηση του κόστου παραγωγής. Για μένα είναι περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Και επίση ποιο θα διαχειριστεί και τα στοιχεία. Η κυρία Χόιμπουχ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ναι, το είπατε και εσείς, ε, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, τίθεται το θέμα ε, της κατοχής των δεδομένων. Ε, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά και στο μέλλον πώς θα γίνεται η διαχείρισή τους. Πολύ συχνά μιλάμε για προσωπικά δεδομένα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, σπίτι μου ε, ε, έχουμε ένα ρομπότ και ο κατασκευαστής έχει πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα. Και πώς θα εκπονούνται οι στατιστικές. Επίσης, είπατε ότι θα πρέπει οι γεωργοί να ασχοληθούν με την τεχνολογία. Ούτως ή άλλως η γεωργία βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία. Κανένα άλλο τομέα ε, δεν έχει βασιστεί τόσο στην τεχνολογία ε, μετά τον πόλεμο όσο η γεωργια βασιζεται σε πολυ μεγαλο βαθμο στην τεχνολογια κανενα αλλο τομεα δεν εχει βασισει τοσο στην τεχνολογια μετα τον πολεμο οσο η γεωργια Το θέμα είναι όμω ποιο θα είναι το κέρδο και τι ασφάλεια προσφέρεται. Δεν δώσατε απάντηση όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων αν ε, στο σπίτι μου χρησιμοποιήσω τη τεχνολογία θα πρέπει να έχω κάποιο πλεονέκτημα. Ε, είτε διευκόλυνση στην εργασία, είτε οικονομική ή ε, εξοικονόμηση χρημάτων. Απλοποίηση της δουλειάς και αυτό δεν καλύφθηκε και αν χρειαζόμαστε κάτι ώστε να παράγουμε πιο εύκολα και πιο οικονομικά. ε, χωρίς να σκεφτόμαστε το κλίμα ή το περιβάλλον, τότε δεν έχει και κανένα νόημα η σύγχρονη τεχνολογία. Θα πρέπει να εξετάσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε, πώς θα το πετύχουμε και θα πρέπει ε, πάντα να κοιτάμε ποιος κερδίζει στην πραγματικότητα. Και όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι οι γεωργοί είναι αυτοί που κερδίζουν από όλη αυτή την υπόθεση. Πολλά πράγματα δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Νόιχλ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα τον ε, μη ρεαλιστικό να θεωρεί κανείς ότι όταν έξω κόσμος εμφανίζει νέες τεχνολογίες και δομές θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε έναν τομέα από αυτές τις νέες δυνατότητες ή ότι, θα, ότι δεν θα προσπαθούσε ένας από τους τομείς της οικονομίας να προσεγγίσει αυτές τις νέες δυνατότητες. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Είχα υπόψη ότι 20% μόνο των γεωργών στην Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης τεχνολογία μέσα από ένα μόνο σημείο εισόδου, στο διαδίκτυο παραδείγματι για τα δεδομένα. Ε, άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή και νέες τεχνολογίες στη γεωργία μόνο για μια πολύ μικρή ομάδα γεωργών. Όλοι οι άλλοι παρακολουθούν τους παραδοσιακούς τρόπους. Γι' αυτούς τι έχετε να πείτε, γιατί κάποια στιγμή είπατε ότι υπάρχει όντως πρόβλημα εάν οι στόχοι της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής είναι και συμπεριλαμβάνουν τη διαφύλαξη της βιοπικιλότητας και βλέπω ότι δεικνύεται. Επομένω, βλέπετε ότι κάποιες μορφές γεωργικής παραγωγής παραδέχεστε πως θα εξαφανιστούν. Το παραδεχόμαστε, γιατί έτσι είναι το ρεαλιστικό. Δεν θέλω λοιπόν αυτό να μου απαντήσετε και επίσης ε, η μικρή κύκλη της αξίας παραγωγής είναι ένας στόχος τον οποίο στο στόχο της βιοπικιλότητας, καλύτερα της πολυμορφίας στη γεωρική παραγωγή θέλουμε να υποστηρίξουμε. Η τεχνολογία, η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα, αλλά μπορεί και να δημιουργεί κάποια άλλα νέα προβλήματα. Επομένω, πώς μπορούμε σε αυτό να δώσουμε απάντηση. Και κάτι άλλο που με ξάφνιασε και πάντα με προξέρει επιφλεκτικότητα όταν μιλούμε για κέρδος αποτελεσματικότητα που σημαίνει συνήθως ε, ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, κάποιων άλλων. Όχι, θα έπρεπε κανονικά να σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε πρωτοπόροι και έρχονται οι άλλοι να μας ακολουθήσουν. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει αναλάβει το ρόλο του, δεν έχει την πρωτοπορία στο χώρο της καινοτομία ε, στην γεωργία, αλλά αυτό που λέμε ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στην παραγωγή μας, στην επεξεργασία και σε αυτό θα ήθελα τη δική σας γνώμη εάν έχει νόημα μακροπρόθεσμα να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα δρόμο για την αποδοτικότητα. Γιατί ναι, μπορεί σε έναν αγώνα δρόμου να βοηθήσουν αυτές οι νέες τεχνολογίες, αλλά δεν δίνουν απαντήσεις σε όρους συστημικούς, παρά μόνο απαντήσεις στο πώς μπορούμε μέσα στο ισχύον σύστημα να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να θέσει το θεμελιώδη ζήτημα τι είδους γεωργία θέλουμε Εάν θέλουμε μια γεωργία προσανατολισμένη προς την παγκόσμια αγορά ή μια γεωργία που να υπηρετεί και να δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με έναν αγώνα δρόμου, ε, μια διελκυστίνδα για την επικράτηση μέσα στο ισχύον σύστημα, ενώ θα έπρεπε να αναζητούμε ένα άλλο σύστημα καταλληλότερα για μας. Ναι, αλλά ε, αν ε, κρατήσουμε απόσταση από τεχνολογίε, τεχνολογίες, δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και κάποια στιγμή θα μας ξεπεράσουν. Ε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και παγκοσμιοποίηση. Οπότε οι, οι πτώσεις είναι παγκόσμιες. Ο κύριος Μπογκόβιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πως ε, με απασχολούν ιδιαίτερα αυτές οι ιδέες. Αυτό που μαζί με τον Σνάρφου Σέν έχουμε ονομάσει ευφυή χωριά, smart villages. Και ναι, δέχομαι ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ψηφιοποίηση, αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η ψηφιοποίηση ενδέχεται να περάσει ξόφαλτσα από τις ε, περιοχές της υπαίθρου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο λοιπόν, η δύναμη έλξη των αστικών κέντρων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και θα αδειάσουν τα χωριά. Γι' αυτό λοιπόν μιλούμε για ευφύ χωριά ως έννοια που προσπαθούμε να εισαγάγουμε σε διάφορου τομείς τη πολιτική, προβάλλοντας αυτό το οποίο και εσεί αναφέρατε, ότι δηλαδή μπορεί να υπάρχουν ακόμα μεγάλε διαφορέ 44% σήμερα μόνο των πολιτών έχουν πρόσβαση σε συστήματα ευρυζωνικότητας και δίκτυα κτλ. Και αυτό θα επιδεινωθεί στο μέλλον. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα επιχειρησιακό μοντέλο στις περιοχές αυτές, της υπαίθρου, που να δίνει λύσεις ένα σύστημα το οποίο να καλύπτεται και από τις κρατικές δομές και σε αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρξει επαρκής συνδεσιμότητα για την Ήπεθρο. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για καλή χρήση των πόρων υδάτινων ε, ή των λοιπασμάτων ακόμη και όλα αυτά που μπορεί να εξυπηρετήσει ψηφιοποίηση, αλλά και οι ανάγκες της ε, σύγχρονης ε, αυτοματοποίησης. αλλά και της ανιχνευσιμότητας. Αυτού δηλαδή που ζητεί όλο και περισσότερο καταναλωτής. Και σε αυτό, αυτό χάρη στην ψηφιακή ε, τεχνολογία μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις και στην ανεχνησιμότητα και σε όλες τις άλλες ανάγκες. Η τεχνολογία αυτή λοιπόν δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη μόνο ή προσβάσιμη μόνο σε ένα μέρος ορισμένους χρήστες. Πρέπει και οι μικρές ή και μεσές εκμεταλλεύσεις να επιτρέπουν στον χρήστη τον καταναλωτή, τον παράγοντα της οικονομίας, την πρόσβαση σε αυτές τις νέες τεχνολογίες ιδάλλως. Θα γίνουμε μάρτυρες της μείωσης των μικρών, του αριθμού των μικρών εκμεταλλεύσεων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τον καταναλωτή. Μια σειρά από εφαρμογές που έχουμε παραδείγματι στην Σλοβενία επιτρέπουν στον καταναλωτή να εξασφαλίσει ανεχνευσιμότητα μέσα από αυτές τις κινητές εφαρμογές που είναι χρήσιμες όχι μόνο για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις αλλά και για τις μικρότερες. Και έτσι πρέπει να εξασφαλίσουμε και την έννοια της κινητικότητας για τις περιοχές της υπαίθρου, καθώς 10% του πληθυσμού τουλάχιστον στην πατρίδα μου μόνο μπορεί να χρησιμοποιεί ε, δωρεάν μεταφορές μαζικές μεταφορές αλλά και η τεχνολογία. Η τεχνολογία χρειάζεται να μπει μέσα σε αυτές τις περιοχές της υπαίθρου. Η τεχνολογία που έχει να κάνει και με την ενέργεια, που έχει να κάνει και με τις αλυσίδες στοιχείων, με τη, το blockchain δηλαδή, και άλλα είναι άλλα κομμάτια του μουσαϊκού που πρέπει να συνδυαστούν για να δώσουμε πάντα το ποιος θα έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες. Γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς και με την αυτοματοποίηση, όπως η στο γάλα, που γίνουν κάποιες ανησυχίες, αλλά και σε άλλους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η αυτοματοποίηση να ε, πείσει, σε αυτό χρειάζεται βέβαια και η ενημέρωση, ώστε να μην χάσουν τον ε, αγώνα αυτών δρόμου οι μικρές εκμεταλλεύσεις, ώστε να παραμείνουν στην, ε, μέσα σε εξελίξεις. Και πρέπει να προβληθούν και οι κοινωνικές πτυχές. Σε αυτό βλέπουμε πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες που δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις εξελίξεις, τις τάσεις. Πρέπει όμως να πείσουμε τον καταναλωτή, φορολογούμενο, πολίτη, ότι μπορεί να υπάρχουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες και μπορούν να τις αξιοποιήσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Υποστηρίζω ιδιαίτερος δε και τη νέα κυνηγερική πολιτική και όλα όσα αυτή περιλαμβάνει σε όρους νέων τεχνολογιών και ό,τι μπορεί να αξιοποιήσει. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσίασή σας. Σχεδόν μας έπεισες. Σχεδόν, λέω. Θα δούμε όμως τι θα μας πει και ο κύριος Δεκάστρο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συνεχίζω στα είπε και ο κύριος Μπόγκοβιτς ότι χρειαζόμαστε τεχνολογία, χρειάζεται οι γεωργοί μας και ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις, το τονίζω αυτό, ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η οργανωτική και εμπορική διάσταση έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία και για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι μικρές και μεσαίες γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις και να έχουν ένα, τη δυνατότητα να παράγουν εισόδημα για τον παραγωγό, χρειάζονται αυτή την ε, τεχνολογία. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα όμως, μια και αναφερθήκατε στον καταναλωτή που απαιτεί όλο και περισσότερο να γνωρίζει ε, τους όρους προέλευσης και παραγωγής του προϊόντος είναι κάτι το οποίο εμείς πάντοτε ζητούσαμε ως κοινοβούλιο, δηλαδή την ενημέρωση για την προέλευση των ε, γεωργικών προϊόντων. Τα συστήματα στα οποία αναφερθήκατε, τα τεχνολογικά, όπως η αλυσίδα στοιχειών, τα blockchain, πώς μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Κατάιναν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι μέλος πολιτικής ομάδας που στηρίζει την καινοτομία. Πιστεύουμε ότι η καινοτομία προσφέρει ευκαιρίες περισσότερο από απειλές. Ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές και τα προβλήματα, αλλά όχι να τα αφήσουμε να εμποδίσουν την πρόοδο. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ήδη χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Υπάρχουν ε, φυσικά μεγάλες διαφορές ε, στα διάφορα μέρη της Ευρώπης ε, και βέβαια κεντρικό είναι το θέμα της διάθεσης ευρυζωνικής σύνδεσης. Μπορεί κανείς να έχει μια εκμετάλλευση που να λειτουργεί με βάση τη διασύνδεση με το διαδίκτυο που έχει στη διάθεσή του. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Θα πρέπει να έχουμε σωστή βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Πολύ συχνά μιλάμε για την προέλευση, για τη συνεργασία παραγωγών και καταναλωτών και για ε, τα μικρά κυκλώματα, αλλά εάν ε, η προέλευση των προϊόντων ε, δεν ενδιαφέρουν ε, όλα τα κράτη-μέλη, εάν μόνο λίγα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται για ηχνηλασιμότητα σε επίπεδο ευρωπαϊκής γεωργικής εκμετάλλευσης, τότε θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ευρώπη. Θα πρέπει όλοι να συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο, να έχουμε ηχνηλασιμότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, Υπάρχει το θέμα των μικρών παραγωγών. Δεν θα πρέπει να τους στρέφουμε τον έναν εναντίον του άλλου. Έχουν καλύτερες, πρέπει να έχουν καλύτερες ευκαιρίε να διαθέσουν στην αγορά τα προϊόντα τους. Μπορεί όμως να υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ιδιοκτησία των δεδομένων. Επίσης, τι ανοιχτά δεδομένα μπορούμε να έχουμε. Πρόκειται για τεχνικά προβλήματα στα οποία θα πρέπει να βρούμε λύση. Πάντως, πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη γιατί λόγω της καθυστέρησης μου δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παρουσίαση της μελέτης. Έχω κάποια σχόλια όμως μετά τις ομιλίες και των συναδέλφων. Και εγώ είμαι υπέρ της καινοτομίας και υπέρ της ψηφιακής οικονομίας. Αλλά θα πρέπει πρώτα να διαρωτηθούμε τι θα εξυπηρετήσει αυτή η ψηφιακή οικονομία και ποιο γεωργικό μοντέλο θα υπηρετήσει. Γιατί αν η καινοτομία και η ψηφιακή οικονομία εξυπηρετούν την ποιότητα των τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία και την κατάκτηση περισσότερων εδαφών, γιατί όχι. Αν η ψηφιακή οικονομία επιτρέψει ε, ανακατάκτηση των εδαφών, την υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Επίσης, αν ασπαστεί την βιώσιμη ανάπτυξη και μια γεωργία που θα σέβεται την απασχόληση και τα εδάφη, γιατί όχι, εμπρός. Αλλά προσοχή, γιατί οι νέες τεχνολογίες έχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν το χάζο μεταξύ των διαφόρων μοντέλων γεωργίας. Και μπορεί να οδηγήσουν σε συγκέντρωση ή υπερσυγκέντρωση, κάτι που είναι αρνητικό. Απ' τη μια λοιπόν χαίρομαι για τις ευκαιρίες που ανοίγονται σε ό,τι φορά την έρευνα και την καινοτομία, αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε και πρώτα να προσδιορίσουμε το μοντέλο που θέλουμε να υπηρετήσουμε τις νέες τεχνολογίες. Και αυτό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε. Θα πρέπει να κάνουμε ένα είδος συγγραφής υποχρεώσεων ε, ή κάποια κριτήρια για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, για να μην παρεκτραπούμε και να μην έχουμε αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή επιδείνωση της σημερινής κατάστασης παρά τις νέες τεχνολογίες ή λόγω των νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε άλλους ε, ομιλητές στον κατάλογο. Οπότε θα ήθελα να κάνω και εγώ λίγα σχόλια. Η η ψηφιακή οικονομία και η ψηφιοποίηση έχει, είναι ήδη πραγματικότητα και έχουν φτάσει και στη Γεωργία. Θα πρέπει όμως να προβλέψουμε και κάποια ρύθμιση αυτών των νέων τεχνολογιών και των φαινομένων. Ε, υπάρχουν όμως κάποιοι κλάδοι και κάποιοι φορείς που δεν ε, ε, είναι υπέρ της ρύθμισης της εξατομίκευσης των δεδομένων της μετάδοσης των πληροφοριών. Γι' αυτό και χρειάζεται ένας αυξημένος ε, έλεγχος και παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας. Να δούμε αν τηρούνται οι προδιαγραφές και τι πρότυπα θα ισχύσουν. Γι' αυτό και σίγουρα χρειάζεται κάποια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό ή σε και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτής της νέας κατάστασης. Αλλά μερικοί δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους ή να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες. Βέβαια θα μου πείτε, γι' αυτό έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Γεωργοί ίσως περιμένουν από εμά να ρυθμίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα τις καλεσμένες μας, Θα δούμε τι θα μας πούν οι εμπειρογνώμονες για όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Σημειώσαμε τις ερωτήσεις. Μάλλον δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις αναλυτικά. Θα ξεκινήσω όμως από την πρώτη ερώτηση. εάν όντως υπερτιμούμε τον αντίκτυπο αυτών των τεχνολογιών ε, στο περιβάλλον, ε, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κλπ. Προσπαθήσαμε στην ε, έκθεση να επισημάνουμε ότι ο πιθανός αντίκτυπος των τεχνολογιών δεν είναι ομαλός, δεν είναι ίσως σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας, ε, σε όλες τις οντότητες ε, της αλυσίδας αξίας υπάρχουν διαφορές που μπορεί να συνδέονται με το μέγεθος, μπορεί να συνδέονται με το είδος της επένδυσης που απαιτείται. Επίσης, όταν μιλάμε για το μέγεθος της εκμετάλλευσης, δεν μιλάμε μόνο για τον αντίκτυπο της επένδυσης, ε, αλλά ε, και της ε, παραγωγής. Το 2010 ο οργανισμός Καλλιλέο διενήρησε μια σειρά δοκιμών που έδειξαν ότι η πλοήγηση η δορυφορική επηρεάζει μόνο γεωργικές εκμεταλλεύσεις από ένα μέγεθος και πάνω. Κάτω από το μέγεθος αυτό το κόστος ήταν υψηλότερο από ότι το όφελος. Δεν λέμε λοιπόν ότι δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν είμαι βέβαιη αν θα πρέπει να μιλάμε για μελέτες. έχουν γίνει δοκιμέ όμως, ε, ιδιαίτερα οι ε, επιχειρήσεις που πολλούν υπηρεσίες ε, που συνδέονται με τις τεχνολογίες αυτές, ε, μετρούν την μείωση της χρήσης νερού, την μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, την αύξηση της παραγωγικότητας. Πρόσφατα, με την συγχώνευση του GNSS και του Κοπέρνικου. Έχουν γίνει και άλλες δοκιμές. Υπάρχουν λοιπόν δεδομένα στην αγορά. Δεν θα μιλούσα για επιστημονικές μελέτες, αυτές καθ' αυτές. Πάντως ε, συνδέονται με τεχνολογίες που βρίσκονται στην αγορά εδώ και κάποιο καιρό. Το GNSS για την πλοήγηση, η δορυφορική πλοήγηση, και ε, οι εξαποστάσεις αισθητήρες είναι δύο από τις ε, τεχνολογίες αυτές. Όταν μιλάμε για το blockchain ή για την ε, τεχνητή νοημοσύνη, βρισκόμαστε στην αρχή των δοκιμών των σχετικών καινοτομιών. Θα δούμε δηλαδή μελέτες για τον αντίκτυπο αυτών στο μέλλον. Δεν είναι λοιπόν ίδια η κατάσταση για όλες τις τεχνολογίες. Ένα στοιχείο που αναφέρεται στην μελέτη είναι η οικονομία του επιμερισμού, η οποία μάλλον θα επιτρέψει και σε μικρές εκμεταλλεύσεις να επωφεληθούν από όλα αυτά. Πάλι βρισκόμαστε σε αρχικό στάδιο της τάσης αυτής. Ε, βλέπουμε όμως κάποια τάση ε, διαμοιρασμού των τρακτέρ, των εφαρμογών Υπάρχουν λοιπόν τρόποι να επωφεληθούν όλοι εξίσου ή σχεδόν εξίσου από τις καινοτομίε αυτές. Ε, κάτι που μάλλον συνδέεται και με κάποιες από τις άλλες ερωτήσεις που τέθηκαν. Πάντως, αυτό που είπατε είναι σωστό και το αναφέραμε. Είπαμε ότι οι γεωργοί δεν μπορούν να φέρουν τον κίνδυνο. χρειάζονται ιδιαίτερα η μικρή παραγωγή χρειάζονται διασφάλιση, πιθανότατα από μεγάλες επιχειρήσεις, από μεγάλες εταιρείε που ε, κάνουν δοκιμές ε, στις τεχνολογίες αυτές. αυτέ. Ε, χρειάζονται λοιπόν κάποιον που να φέρει το κόστος και τον κίνδυνο Προφανώ θα πρέπει να γίνουν διάφορε δοκιμέ ε, προτού φτάσουμε στο σημείο όπου η χρήση των τεχνολογιών αυτών θα ε, επιφέρει αποκλειστικά ωφέλη και όχι τον ε, κίνδυνο λαθών. Αυτό το σενάριο ισχύει για όλες τις τεχνολογίες. Όπως όμως έχει αναφερθεί και πριν, δεν θα σταματήσει να εξελίσσεται η τεχνολογία υπάρχουν μεγάλοι παράγοντες, υπάρχουν μεγάλοι μη ευρωπαϊκοί φορείς που επενδύουν πολλά στις τεχνολογίες αυτές και θα τις διαθέσουν στην αγορά και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που ε, θα έχουμε ε, όξυνση της κατάστασης όσον αφορά τα μονοπόλια, όπως αναφέρθηκε και πριν. Uh, Θέλω να συνεχίσω και εγώ σε αυτό την απάντηση, γιατί στη μελέτη ε, δεν, δεν, κάναμε προσέγγιση επιλογής υπέρ ή κατά της ψηφιοποίησης. Κοιτάξαμε να καταγράψουμε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο με την πρόοδο της ε, τεχνολογίας και τα τεράστια ωφέλη που αυτή φέρνει. Όπως είπε και η Μόνικα νωρίτερα, έχουμε ήδη μεγάλες, τεράστιες πολυεθνικές που υποστηρίζουν αυτές τις εξελίξεις τεχνολογία. Ξέρουμε μόνο ότι όποιος συμμετέχει κερδίζει και σε όρους εισοδήματος και σε όρους ανταγωνιστικότητας και η πρόκληση είναι να δούμε πώς οι λοιποί στόχοι των κοινωνιών μας, δηλαδή περιβάλλον, κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, κλιματική αλλαγή, πώς και αυτοί οι τομείς μπορούν να ωφεληθούν από τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Το αν είναι θετική ή όχι, η εξέλιξη της δεν είναι δικό μας θέμα, δεν είναι κάτι που εμείς θα κρίνουμε. Απλώς προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όλους τους στόχους, έτσι ώστε να ωφεληθούν με τις νέες δυνατότητες από αυτές τις εξελίξεις. Στη μελέτη μιλούμε για τους συνεταιρισμούς και τις προκλήσεις που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν και λέμε ότι ίσως με τους συνεταιρισμούς μπορούμε να έχουμε ένα παράγοντα ε, διάχυσης της γνώσης, αντιμετώπιση των προκλήσεων και για το ύπεθρο και για το περιβάλλον με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, ως διαμεσολαβητές δηλαδή γνώσεων. Αν θες και να πεις κάτι, για να συμπληρώσω στο θέμα αυτό. Ο στόχος της μελέτης είναι να έχουμε μια ε, γενική επισκόπηση από ψηλά των ε, εξελίξεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λύνονται όλα τα προβλήματα της γεωργίας, προφανώς. Τα πλεονεκτήματα σε όρους περιβάλλοντος, χρήση λιπασμάτων, ε, υδάτων κτλ. Με την έρευνα της τεχνολογίας, αλλά και με το ίντερνετ των πραγμάτων, το έδεικτο των πραγμάτων βοηθά ε, χάρη στην ε, παρακολούθηση και την ε, καταγραφή της πορείας προληπτικά, δηλαδή μπορεί να μας εξασφαλίσει μια στοχευμένη χρήση αντί να χρησιμοποιούμε τα λοιπάσματα για να προλαμβάνουμε τις ασθένειες μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν έχουν ανοιχνευτεί αυτές ή με μια πιο ευφύη χρήση των πόρων. Κατά κάποιον τρόπο με τη νέα τεχνολογία μπορούμε να αντιστρέψουμε τον τρόπο χρήσης των πόρων αυτών ή των λοιπασμάτων, αντί να είναι προληπτικός, να είναι μόνο όπου υπάρχει ανάγκη. Απάξει και διαγνωστή ανάγκη. Με στόχο όχι πάντα και μόνο την αύξηση παραγωγής, γιατί αν είναι ευφιέστερη η παραγωγή, πάλι ο γεωργός θα έχει μεγαλύτερο κέρδος ή μεγαλύτερο περιθώριο. Με σταθερή παραγωγή δηλαδή και ευφυή παραγωγή θα έχει μεγαλύτερο περιθώριο. Ένα άλλο στοιχείο που έχει μεγάλη σημασία, είναι κρίσιμο και είναι δύσκολο να το αναλύσουμε, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι το πώς η τεχνολογία μπορεί και οφείλει να αλλάξει τις γεωργικές πρακτικές. Και στην πράξη, όταν, μιλούμε, όταν συνομιλούμε με τους γεωργούς, νιώθουμε ότι είναι αγχωμένοι από το γεγονός ότι πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο μπροστά σε έναν υπολογιστή και να προσπαθήσουν να αναλύσουν στοιχεία, κάνοντας κάτι που δεν είναι δική τους δουλειά. Εκείνοι θέλουν να βρίσκονται στο αγρόκτημα. Θέλουν ε, να ασκούν την γεωργική τους δραστηριότητα. Οπότε μια πρόκληση είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες με τρόπο που οι γεωργοί θα λαμβάνουν μόνο τις χρήσιμες για αυτούς πληροφορίες για να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Για να μην του αναγκάσουμε ε, ή να απαιτούμε να γίνουν ε, εμπειρογνώμονες για κάτι που δεν είναι δουλειά τους. Ούτε θα πρέπει να ασχολούνται αυτοί με την ανάλυση των μαζικών δεδομένων. Και αυτό θα επηρεάσει την αλυσίδα αξιών. Και σίγουρα οι επιχειρήσει επιχειρήσεις ε, γίνονται τμήμα και οι αγροτεχνολογικές επιχειρήσει γίνονται τμήμα τη αλυσίδα αξιών. Γιατί δεν μπορούν οι γεωργοί να γίνουν αναλυτέ δεδομένων ή να χειρίζονται μαζικά δεδομένα. Θέλουν κάποιες πληροφορίες μόνο για να λαμβάνουν περιστατωμένα τις αποφάσεις τους όταν χρειάζεται να λάβουν αποφάσεις. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε, να δούμε εδώ τι αντιστάθμισμα θα βρούμε, τι αντάλλαγμα θα δοθούν, στο πώς ε, ε, οι ρηξικέλευτες αυτές τις τεχνολογίες επηρεάζουν την αλυσίδα αξιών. Θα πρέπει να αλλάξει η αλυσίδα αξιών, αλλά όχι ε, να αλλοιώσει και το, το βασικό χαρακτήρα, την πεμπτουσία του Γεωργού, γιατί ο Γεωργός θα πρέπει να επικουρείται στην γεωργική του δραστηριότητα με τις νέες τεχνολογίες, αλλά παρόλα αυτά να κρατά τη βασική του γεωργική δραστηριότητα που είναι δουλειά στο αγρόκτημα. Και αυτός ο συμβιβασμό θα είναι σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Τώρα, η ιδιοκτησία των δεδομένων. Ποιος είναι ο κύριος των δεδομένων. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά προς το παρόν ε, μένει αναπάντητο το ερώτημα της κυριότητας των δεδομένων και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Η αγορά πάντως δεν δίνει ακόμη μία απάντηση, γιατί η δική μας μελέτη ανάλυσε την, τον αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογιών στην αλυσίδα αξιών. Ήρθαμε φυσικά σε επαφή με πολλούς κρίκους αυτής της αλυσίδας αξιών, ανάλογα με το συνομιλητή μας η απάντηση είναι διαφορετική. Γιατί ναι, μεν τα δεδομένα είναι ευαίσθητα, αλλά τα δεδομένα μερικές φορές είναι και αγαθό, είναι οικονομικό στοιχείο. Ε, και η ιδιοκτησία των δεδομένων σημαίνει μέγεθος επιχείρησης και η ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να μην ικανοποιεί όλους τους φορείς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη γεωργία, ισχύει και για άλλους ε, κλάδους που περνάνε από την ίδια διαδικασία ψηφιοποίησης. Οπότε η συζήτηση είναι ευρύτατη, αλλά νομίζω ότι είναι αμυγός πολιτική, πολιτικού χαρακτήρα. Και δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση. Μία και μοναδική απάντηση μπορούν να δώσουν εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά, τεχνοκράτες. Όσον αφορά το θέμα των δεδομένων, η μελέτη μας κάνει τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε διάφορα είδη δεδομένων και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν διάφορα είδη δεδομένων, άρα θα πρέπει να τα χειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν δεδομένα που προέρχονται από τα μηχανήματα, καθαρά τεχνικά δεδομένα δηλαδή, ενώ έχουμε και δεδομένα που, όπως είπατε, είναι προσωπικά δεδομένα όπου ισχύει ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Όσον αφορά τον τομέα ή το κάθε πρόσωπο θα ισχύει πάντα η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε και όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι αισθητήρε και οι νέες τεχνολογίες. Όχι μόνο η πρόσβαση σε αυτά, αλλά και ο τρόπος που συλλέγονται και αποθηκεύονται είναι κάτι σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Θα ήθελα να, να προσθέσω κάτι για τα δεδομένα. Όσον αφορά το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το ίντερνετ ε, στη γεωργική εκμετάλλευση, ε, συχνά αναφέρεται η υποδομή, οι υποδομές πληροφοριών, ε, και δεν είναι απαραίτητο να ε, ε, μοιραζόμαστε τις ίδιες τεχνολογίες, γιατί αυτό μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα. Όσον αφορά το blockchain, που συζητιέται πάρα πολύ, την ε, αλυσίδα συστοιχιών, πρόκειται για ένα μητρό συναλλαγών, το οποίο σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβαίνει, καταχωρίζεται χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η διαφάνεια. Μπορεί κανείς να βρει την πηγή των προβλημάτων και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για στόχους που συνδέονται με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος. Ε, μπορεί να έχει κανείς στοιχεία για το σύνολο της ε, αλυσίδας ε, αξίας και μπορεί αυτό να αυξήσει την εμπιστοσύνη των γεωργών. Θεωρούμε ότι είναι μετρίου αντικτύπου η τεχνολογία αυτή. Υπάρχουν διάφορες σχετικές μελέτες. Δεν πιστεύουμε όμως ότι αμέσως θα έχει τεράστιο αντίκτυπο. Νομίζω όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα, ότι αξίζει να παρακολουθούμε στο μέλλον. Η κυρία Κύροβα, όσον αφορά το blockchain υπάρχουν δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι είναι αποκεντρωμένη τεχνολογία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αρχή, κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο ε, που να το διέπει και το δεύτερο είναι ότι είναι ασφαλές επειδή είναι κρυπτογραφημένες όλες οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένα τα δεδομένα ανάμεσα στον αποστολέα και τον αποδέκτη. και δεν μπορεί κανείς να διαγράψει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες από τη στιγμή που έχουν καταχωριστεί. Γι' αυτό, από τη στιγμή που έχουν μπει στην αλυσίδα, δεν μπορούν να τροποποιηθούν από κάποιο πρόσωπο ή κάποιον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι πριν δύο ή τρία χρόνια είχαμε μία περίπτωση αυγών μολυσμένων ε, στην ε, Γαλλία και δεν γνωρίζαμε πού ακριβώς ξεκίνησε το πρόβλημα. Ούτε γνωρίζαμε ποιοι είχαν ε, λάβει τα προβληματικά αυγά. Σε μια τέτοια περίπτωση η τεχνολογία blockchain, όπου καταχωρίζονται οι πληροφορίες με ασφαλή τρόπο και ε, ε, διαβιβάζονται σε όλους ε, τους ενδιαφερόμενους, μπορεί κανείς εύκολα να αντιμετωπίσει που υπήρξε το πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα αξίας και μπορεί να διαπιστώσει ποιοι προμηθευτές έχουν επηρεαστεί, έχουν λάβει τα προβληματικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Μια και δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Σας έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο για τις απαντήσεις. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και σίγουρα η μετάδοση των πληροφοριών και η διευκόλυνση αυτής της μετάδοσης των πληροφοριών ε, απαιτείται στον τομέα αυτό, θα είναι πολύ χρήσιμη και απαραίτητο στοιχείο της πρόοδου και της καινοτομίας. Ο Γιώργο, όμω, από τη στιγμή που καλείται να λάβει κάποιε αποφάσει, θα πρέπει να κάνει προηγουμένω ε, κάποια ανάλυση. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε ίσω μεθοδολογικά κάποια στοιχεία, κάποιε στατιστικές πληροφορίε για να τον βοηθήσουμε. Αλλά την απόφαση τελική ανάλυση θα τη λάβει ατομικά ο Γεωργός. Γιατί αυτό γνωρίζει το χωράφι του, αυτός γνωρίζει το ζωικό του κεφάλαιο και ξέρει πώ θα τα διαχειριστεί. Αυτή είναι η δουλειά του αγρότη, Γιώργου ή κτηνοτρόφου. Και μερικές φορές βέβαια κοιτάν την κατάσταση του αγροτεμαχίου ή του κοπαδιού στην ε, οθόνη, αλλά σίγουρα η και μερικες φορες βεβαια κοιταν την επιτόπου είναι η πιο σημαντική. Αλλά είναι σημαντικές όλες αυτές οι τεχνολογίες ε, και ειδικά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά για την μελέτη που εκπονήσατε. Βλέπετε ότι προκάλεσε πολλές απορίες και πιστεύω ότι θα περάσουμε σε μια νέα φάση με όλες αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά τεχνικό διάλειμμα για να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Περνάμε στο επόμενο σημείο της της διάταξή μα. Θα ήθελα να καλωσορίσω του καλεσμένου μα Το σημείο αυτό αφορά τη δημόσια ακρόαση με θέμα τις εξελίξεις στο πλαίσιο επιδόσεων τη κοινή γεωργική πολιτική. Η δημόσια αυτή ακρόαση εμπίπτει στο τρέχον κοινοβουλευτικό μας έργο για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ε, μεταβαίνουμε προς μια κοινή γεωρική πολιτική που θα στρέφεται περισσότερο προς τι επιδόσεις, κάτι που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του, της θέσμης μεταρρυθμίσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος λοιπόν αυτής της σημερινής δημόσιας ακρόασης είναι μια αξιολόγηση και η ανάλυση του τρέχοντος ε, κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης και η εξέταση όλων αυτών στο πλαίσιο ε, της, των εξελίξεων ε, του νέου νομοθετικού πακέτου. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους καλεσμένους εμπειρογνώμονές μας που είχαν την καλοσύνη ε, να λάβουν μέρος στη δημόσια κρόση και να μας παρουσιάσουν τις αναλύσεις και τις απόψεις τους στον τομέα αυτό και να περάσουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή στην παρουσίαση των εκθέσεων των εμπειρογνώμονων μας. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Αντώνιο Λιμόνε, που είναι Γενικός Διευθυντής του Πειραματικού Ινστιτούτου Προλήψης των Ζωονόσων του Μετζοτζόρνο. Κατόπιν θα λάβει το λόγο ο κύριος Βαυζίνης Τσούμπακ, που είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πόσναν στις επιστήμες της ζωής, ε, τμήμα οικονομικών και οικονομικής πολιτικής της αγροτικής οικονομίας. Και τρίτος, το λόγο θα έχει ο κύριος Ιβ Μάντρα, που είναι πρόεδρος ε, και συντονιστής στο Farm Europe. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Οι καλεσμένοι μας έχουν από ένα δεκάλεπτο καθένας και θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Αντώνιο Λιμόνε Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Λιμόνε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο το όνομά μου. Το μικρόφωνο του μιλητή έχει κλείσει. Το μικρόφωνο του μιλητή, παρακαλώ. Ξεραρχίστε, παρακαλώ, λέει ο πρόεδρος. Προέρχομαι λοιπόν από την Καμπανία. Το Ινστιτούτο που εκπροσωπώ εγώ έχει ιστορία 200 ετών. Ασχολείται με την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι οργανισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης που μεριμνά για την ασφάλεια των τροφίμων προς όφελος του πολίτη. Και ξεκινώ με αυτούς τους στόχους όπως τους ορίσαμε εμείς στην καμπανία μέσα από τρία σκέλη οργάνωσης καινοτομία και ενημέρωση αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που μας δείχνουν ότι είναι πιο νέοι τώρα οι γεωργοί, όχι μόνο στο νότο της Ιταλίας και την Καμπανία ειδικότερα, αλλά σε όλη την Ιταλία. Έχουμε τον, το σκέλος της πράσινης ε, καμπανίας με τη βιώσιμη γεωργία, την προστασία και αξιοποίηση των γεωργικών περιοχών, την βελτίωση των επιδόσεων σχέση με το περιβάλλον δεδομένων των συνθήκων και των πολιτικών μας στόχων και η αλληλέγγυα καμπανία η οποία στοχεύει στην ποιότητα ζωής και απόλαυση των ωφελών για όλους. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ε, μοντέλο εδαφικής οργάνωσης που λαμβάνει υπόψη και τις διαφορές που επικρατούν στην περιφέρειά μας, γιατί δεν είναι ομοιογενής, έχει πολύ μεγάλες διαφορές από μια περιοχή στην άλλη. Έχουμε δύσκολη γεωγραφία και αυτό το λέω γιατί μπορεί λόγω της ιδιαιτερότητας και της ε, πληθώρας βιοπικιλότητας που γνωρίζουμε να οδηγηθούμε σε προβλήματα ως προς την υλοποίηση και απόλαυση των ωφελών της νέας ΚΑΠ σε ένα τόσο ποικίλο περιβάλλον και έδαφος. Δεν ε, μπορώ να πω βέβαια ότι έχουμε κακά αποτελέσματα. Μάλλον έχουμε μπορέσει να καταγράψουμε πολύ θετικέ επιδόσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 με βάση παραμέτρους που είχαν οριστεί, τις οποίες έχουμε σε ένα βαθμό ξεπεράσει, σε κάποιες άλλες πολυπόμεθα, άρα έχουμε και αρκετή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Ωστόσο, το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγηση πάνω στο οποίο στηρίζεται η νέα ΚΑΠ 1420 ε, περιγράφει κάποιες υποχρεώσεις αξιολόγησης. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν που έχουμε φτάσει εμείς με το πλαίσιό μας αυτή τη στιγμή, πλάσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, που στηρίζεται σε δύο στοιχεία. Ένα ενιαίο για κάθε κράτος και άλλο ένα όπου το output του κάθε κράτους μέλους πρέπει να ε, περιγραφή και να αναγνωστεί πιο συγκεκριμένα με βάση τους στόχους που θα έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων σε τοπικό, περιφερειακό δηλαδή ή εθνικό επίπεδο. Μέσα από αυτό το σύστημα λοιπόν εμείς περιγράψαμε την κατάσταση διαγνώσκοντας ε, τα όρια με, τα, με τους τέσσερις δείκτες συστημικό ανταπόκριση αποτελέσματος ε, και επιπτώσεων ή αντικτύπου που θέλουμε να παρακολουθούμε και τους περιορισμούς ή τις δυσκολίες που έχουμε στην καταγραφή των αποτελεσμάτων και λόγω των διαφορών ενδιαμέσων, άρα χρειάζεται μια απλοποίηση, ε, χρειάζεται ένα πλαίσιο επιδόσεων το οποίο να επιτρέπει και την ετήσια αξιολόγηση η παρακολούθηση, η δυσκολία που βλέπουμε να, να γνωρίσουν και άλλες περιφέρειες Ιταλίας. Ε, που επιβραδύνουν ουσιαστικά το σύστημα και την ε, αξιολόγηση και τη λειτουργία των προγραμμάτων. Άρα μέσα σε ένα χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει το πρόγραμμα να είναι πιο μακροπρόθεσμο γιατί είναι πολύ στενά τα όρια τα χρονικά το ετήσια για την αξιολόγηση. Και έτσι προχωρώντας προς τη νέα ΚΑΠ και τους στόχους παρακολούθησης για την περίοδο 2021-2027 και αξιολόγηση αντίστοιχα. Οι στόχοι της αξιολόγησης, επομένως είτε οι επιδόσεις, προσδορισμός των παρεμβάσεων, είτε η υπευθυνότητα αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και η αποδοτικότητα σχέση με την ποιότητα των παρεμβάσεων, αλλά και η διαφάνεια σε σχέση με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, σημαίνουν ότι η παρακολούθηση αυτή θα έχει οριστεί με βάση κάποιες προόδους για την υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών και θα έχει δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν εκεί βεβαίως η δαπάνη θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά πάλι και αυτό με κάποια όρια ως, δείκτης, ως σημείο αξιολόγησης. Αυτό που βλέπουμε σαν πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει απλοποίηση στο σύστημα προσμέτρησης των επιδόσεων, δηλαδή βλέπουμε κίνδυνο από τη συγκεκριμένη δυνατότητα να καταστεί πολύ περίπλοκο το σύστημα μέτρησης ε, το, της στήριξης των στόχων, ενώ κανονικά ο στόχος μας είναι η απλοποίηση. Και αυτό που λέμε πάντα είναι απλοποιούμε, απλοποιούμε, αλλά τελικά αυτό δεν πραγματοποιείται. Έτσι λοιπόν έχουμε δείκτες όχι μόνο δαπανών, αλλά και παραγωγής και αποτελέσματος και αντικτύπου. Και έτσι φαίνεται πολύ πιο σημαντικό και επαχθές και φιλόδοξο αυτό το εγχείρημα. Πολύ πιο περίπλοκο λοιπόν. Ίσως όμως μπορεί το ε, μοντέλο αυτό της περιφερειακής ανάπτυξης μέσα στην ΑΠ να αποδειχθεί τελικά περιορισμένης ε, αποδόσεις. Είναι πολλές λοιπόν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, οι δημόσιες αρχές στην Ιταλία, είτε κεντρικό κράτος είτε περιφερειακές αρχές. Και άρα υπάρχουν αμφιβολίες στο κατά πόσο είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε μια απλοποιημένη ΠΑΚ με αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης ε, που επιβάλλονται και που είναι περίπλοκα και επαναληπτικά πολλές φορές. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε μια δομή που θα κρίνουν οι Βρυξέλλες, μια δομή όμως που μένει πολλά χιλιόμετρα μακριά, που βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τις Βρυξέλλες και θα πρέπει να αξιολογηθεί με έναν τρόπο αρκετά περίπλοκο. Πολύ δύσκολο αυτό. Ξέρουμε ότι η τέχνη της πολιτικής είναι τέχνη περίπλοκη, τέχνη δύσκολη. Αλλά πολλά θα κρυθούν από τις προσπάθειες, από τις επιλογές που θα μπορούσαν να είναι παραδείγματι τα πιο σημαντικά και αξιόλογα στοιχεία της ΚΑΠ να μπουν μέσα σε ένα σύστημα στήριξης πολύ πιο στοχευμένος με βάση αποτελέσματα αλλά και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να λησμονούμε πω όταν κάποιο ε, ζητεί ένα πρόγραμμα, επιβάλλει ένα πρόγραμμα ή προτείνει ένα πρόγραμμα, πρέπει και να καλείται να το τηρήσει. Δηλαδή, εννοείται ότι αν κάποιο δίνει χρήματα για ένα πρόγραμμα, θα περιμένει και να τηρηθούν οι όροι του προγράμματο στην περιφέρεια ενδεχομένω τη Ευρώπη. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα βλέμμα προ την αποδοτικότητα τη δράση, ναι, αλλά και μια αξιολόγηση του εάν αυτοί οι δείκτε output αποδοτικότητα είναι ανεξέλεγκτη δηλαδή και ξέρουμε βεβαίως ότι δεν ε, μπορούν να λειτουργήσουν ε, όλα τα εγχειρήματα και τα έργα με βάση την περιφερειακή δομή αλλά πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους με αξιολόγηση και επαλήθευση των επιλογών. Άρα λοιπόν θα ήταν ίσως ε, σκόπιμο να γίνει μια επιλογή και ανάγνωση ενδεχομένως του κατά πόσον τα αποτελέσματα υλοποιούν τους επιδοχθέντες στόχους, αφήνοντας όμως και ένα περιθώριο πρωτοβουλίας στην ε, τοπική οργάνωση, τοπική δομή, με τα όρια βεβαίως που θα θεωρηθούν ε, σκόπιμα. Περίπλοκο λοιπόν όλο αυτό και σε σχέση με την πράσινη οικονομία θα ήταν, ε, πιστεύω, σκόπιμο ιδιαίτερος να εντοπιστούν συγκεκριμένοι δείκτες για το κλίμα, το περιβάλλον, που να λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες για ε, όλους τους γεωργούς ή και ιδιαίτερα για τις πιο περιθωριακές όπως ονομάζονται περιοχές να μεταβούν, να εξασφαλίσουν τη μετάβαση μέσα σε ένα νέο μοντέλο ένα μοντέλο το οποίο ταυτόχρονα θα ε, στηρίζει, θα ανταμείβει τις ε, εκμεταλλεύσεις εκείνες οι οποίες κάνουν καλύτερη δουλειά και τηρούν τις προϋποθέσεις. Και έτσι αναφέρομαι σε μια νέα ΠΑΚ 21-27 με ένα σύστημα στηριγμένο σε επιδόσεις ναι και στα αποτελέσματα, αλλά που ταυτόχρονα θα μπορεί μέσα από τα στρατηγικά έργα να εντοπίζει την ανάγνωση, την ορθή ανάγνωση των αποτελεσμάτων και ξέρω ότι στις περιοχές αυτές και ιδιαίτερα τη δική μου, την καμπανία είναι δύσκολο να αναγνωστούν σωστά τα αποτελέσματα γιατί υπάρχουν στοιχεία στην πραγματικότητα, στην πράξη τη γεωργική και την κτηνοτροφική στην περιοχή μου, ιδιαίτερα στην ε, κτηνοτροφία που έχει πανάρχες ρίζες. Από τον 7ο αιώνα π.Χ. όταν έγραφε την Οδύσσια ο Όμηρος, ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο βοσκός κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που έκανε και ο βοσκός την εποχή του Οδυσσέα. Άρα λοιπόν όταν ζητούμε παράγοντες καινοτομία σε μια τέτοιου είδους οικονομία, και εδώ είναι η έκκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι χρειάζεται ένα, μια περιοχή που έχει διαρθρώσει περίπλοκη και δομές πολυσχηδείς, να αναγυγνώσκεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην χαθεί το τελικό ε, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και να μην φτάνει τελικά το ράσο να κάνει τον παπά. Ιδιαίτερα αν το ράσο έχει γίνει στενός κορσές. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε εάν οι στόχοι που έχουν προσδοριστεί εκ των προτέρων είναι πράγματι οι κατάλληλοι και για να μπορέσουμε να διαβάσουμε σωστά το σύστημα πρέπει και να δώσουμε εμπιστοσύνη στους, ε, στις τοπικές αρχές και δομές με προσοχή, με ευθεία κτλ. Αλλά και με πολύ μεγάλη προσοχή και επιφυλακτικότητα να διαθέσουμε τους σπόρους που χρειάζονται, ώστε να μην διασπαθιστούν βεβαίως, αλλά και ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η Ευρώπη, η χρήσιμη, η ευεργετική, για ένα περιβάλλον για μια περιφέρεια η οποία και διαφυλάσσει το χαρακτήρα της υπαίθρου, της τοπικής οικονομίας, ενός συστήματος και μιας οικονομίας που η Ευρώπη πρέπει να, να αξιοποιεί, να αναδεικνύει και όχι να υπονομεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στον επόμενο μας καλεσμένο τον καθηγητή Τσούμπακ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καταρχήν είμαι οικονομολόγος. Δεν εργάζομαι στην διοίκηση, αλλά μια και μιλούμε για μια στροφή της κοινή γεωργικής πολιτικής προς τα αποτελέσματα, προς τις επιδόσεις, θα σας δώσω κάποια αποτελέσματα που είναι αποτελέσματα της κοινή γεωργικής πολιτικής όπως έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Ε, είμαι Πολωνός, γι' αυτό και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της κοινή γεωργικής πολιτικής, κυρίως στην Πολωνία. Ε, θα ήθελα εν συντομία να σας ε, αναφέρω τέσσερις βασικούς τομείς. Να μιλάω πιο αργά, μάλιστα. Εντάξει, λίγο πιο αργά θα μιλάω για να προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, την ε, στήριξη, την ενίσχυση και την απόφαση για τον ορισμό του πραγματικού γεωργού. Επανερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση για τον ορισμό του γεωργού. Ε, γίνεται μια απόπειρα του ορισμού του τι είστε σήμερα αγρότης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο ε, στηρίζεται κυρίως στην οικογενειακή εκμετάλλευση. Σε αυτό το μοντέλο οικογενειακής ε, γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τα βασικά, τρία βασικά κριτήρια που βλέπετε στην αρχή. Καταρχήν, έχουμε μεμονωμένες ατομικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, λαμβάνεται υπόψη βέβαια και η οικογένεια, δεν είναι μόνο ατομική, είναι συνήθω οικογενειακή η εκμετάλλευση, αλλά το 50% του εργατικού δυναμικού είναι κυρίως προσωπική εργασία ή η εργασία των μελών της οικογένεια. Και υπάρχει και ένα οικονομικό κριτήριο, γιατί όπω είπα είμαι οικονομολόγο, και ε, σίγουρα και η Γεωργία ε, έχει και οικονομικά αποτελέσματα. Μιλούμε για αγροτική οικονομία. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη το κατά κεφαλήν ε, εισόδημα που είναι υψηλότερο από το κατώτατο ε, μισθό σε άλλους τομείς. Έχουμε περίπου 12 εκατομμύρια, πάνω από 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις και είναι λιγότερο από 10% ε, της τυπικής απόδοσης. Και αυτό το λέμε χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Ουσιαστικά έχουμε μόνο πέντε με βάση το FADN γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με βάση αυτό το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Και την ελάχιστη, το, το κατώτατο μισθό το, ε, τον λαμβάνω περίπου ένα εκατομμύριο. Ενώ έχουμε ε, 4 εκατομμύρια φάρμες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις με ε, εισόδημα πάνω από το καθαρό κατώτατο, αλλά έχουμε και ε, 3 περίπου εκατομμύρια οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, ενώ περίπου 360.000 μεγάλης ε, κλίμακος εμπορικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, και οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις είναι περίπου το 30% ε, του συνολικού αριθμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, 4 εκατομμύρια λαμβάνουν περίπου το μέσο μισθό, ενώ περίπου μισό εκατομμύριο είναι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν αυτό το μέσο μισθό και είναι 5% του συνολικού αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 5% είναι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και ε, παράγουν το 20% της συνολικής αξίας της παραγωγής. Εδώ έχουμε το καταμερισμό αναχώρα σε ό,τι αφορά την κόκκινη στήλη, ε, που αφορά τις ε, μεγάλες εταιρείες, μεγάλες κλίμακος ε, εμπορικές εταιρείες, έχουν περισσότερους απασχολούμενους, αλλά είναι πολύ μικρό το μερίδιό τους στην παραγωγή. Οπότε η αποτελεσματικότητα της γεωργικής εργασίας ε, είναι σίγουρα μεγαλύτερη στις ε, μεγάλες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Παρόλο που είναι μικρός ο αριθμός τους, είναι μεγάλο το τμήμα της τυπικής τους απόδοσης. Για να δούμε τώρα τα αποτελέσματα τη κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πιο πρόσφαρε συνθήκε για φιλοπεριβαλλοντικέ επενδύσει. Εδώ έκανα ένα μοντέλο για την Πολωνία χρησιμοποιώντα τα στοιχεία από το 1993 μέχρι το 2004. Βλέπετε τις κόκκινες στήλες που δείχνουν το μοντέλο που θα ίσχυε στην, Γεωργία, δεν είχαμε, στην Πολωνία δεν είχαμε την κοινή γεωργική πολιτική. Και επίση έχουμε τις επενδύσεις ε, για τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Και βλέπουμε ότι η καθαρή αξία ε, των επενδυτικών δαπανών και κυρίως μετά το 2004 είναι πολύ μεγαλύτερες, περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. που είναι τα συνολικά ωφέλη από την ε, αρχή της ένταξης της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε μεγάλη αύξηση στις ε, γεωργικές επενδύσεις στην Πολωνία μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ένα ε, μεγάλο τμήμα αυτών των επενδύσεων είναι επενδύσεις στην καινοτομία. Επίσης, έχουμε κάποια στοιχεία για τον γεωργοτροφημικό τομέα, που επίσης ε, συγκέντρωσε των επενδύσεων. Πάντως, ε, είναι μεγάλη η προσθέμενη αξία της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής και στην Πολωνία. Και βλέπετε πόσο ανθεκτικές είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Το 2008 και το 2009, παρά την κρίση γιατί ήταν ε, βαθύτατη κρίση και επηρέασε κυρίως τις επενδύσεις ε, στον αγροδιατροφικό κλάδο, αλλά παρόλα αυτά, σε σχέση με άλλους τομείς, υπήρξε μια ανθεκτικότητα της γεωργίας. Και αυτό χάρη στον μηχανισμό με τον οποίο φτάνουν οι, οι ενισχύσεις της επενδύσης της γεωργίας σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη ελαστικότητα του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, εδώ να σας περιγράψω με συντομία την μεθοδολογία. Καταρχήν λάβαμε υπόψη όλες τις δραστηριότητες του δεύτερου πυλώνα, ανάλογα με το τι εξυπηρετούν. Αν δηλαδή εξυπηρετούν ένα βιομηχανικό γεωργικό μοντέλο, ε, αν εξυπηρετούν το μοντέλο μιας κοινωνικά βιώσιμης γεωργίας ή μια, ε, μιας φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας. Σε ό,τι αφορά την Πολωνία, όπως σας είπα, χρησιμοποιήσαμε πολύ διαφορετικά κριτήρια από ότι το διοικητικό καταμερισμό. Σε ό,τι αφορά το, τους... Ε, εμείς κάναμε τη διάκριση μεταξύ των δικαιούχων, δηλαδή αν ήταν ε, ε η ύπεθρος ή ιδιοκτήτες ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δασών και αγροδιατροφικός κλάδος ή ε, αν ο στόχος ήταν η ενίσχυση, ανάλογα με, την, ε, με το κεφάλαιο ε, και με το ποια στοιχεία του ενεργητικού λάβανε τις ενισχύσεις. Και κάναμε τη, ανάλυση, τη στατιστική ανάλυση για όλες τις χώρες και τις ομαδοποιήσαμε σε τρεις κυρίως ομάδες. Θα σας δείξω τα αποτελέσματα των τριών αυτών ομάδων και τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Η πρώτη ομάδα είναι η Δανία, η Ιρλανδία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες αυτές ε, που είναι το 60% του δεύτερου πυλώνα για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, το 60% των πόρων ε, δόθηκαν σε περιβαλλοντικές δράσεις. Και οι χώρες αυτές ε, έκαναν πολύ περισσότερες επενδύσεις στις ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και επίσης υπήρχε μία ισορροπία μεταξύ των ε, γενικών γεωργικών επενδύσεων και των ειδικών περιβαλλοντικών γεωργικών επενδύσεων. Και επίσης, αν δούμε το μέσο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης, βλέπουμε ότι η πρώτη ομάδα αυτή, η φιλοπεριβαλλοντική, είναι η μεγαλύτερη και εκεί είχαμε λιγότερη απασχόληση εργατικού δυναμικού, αλλά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στη γεωργία. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων. Έχουμε πολύ καλύτερη εξισορρόπηση του γεωργικού και του περιβαλλοντικού στοιχείου. Και αυτό είναι σημαντικό τμήμα της συζήτησης, ε, ο περιβάλλοντος και γεωργίας. Και έρχομαι εδώ στα συμπεράσματα. το ύψος των δαπανών ε, ανταποκρίνεται στο, στο βαθμό ανάπτυξης μιας χώρας. Όσο πιο ανεπτυγμένη είναι μια χώρα, τόσο περισσότερες ε, δαπάνες κάνει ε, για τον περιβάλλον, σε ό,τι αφορά τις προαιρετικές ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα, δηλαδή τις περιβαλλοντικές. Και φυσικά υπάρχει διαφορά μεταξύ των παλαιότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πιο νέων χωρών οι παλαιότερες χώρες έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα και μεγαλύτερη υποστήριξη. Και εδώ έχω μερικά στοιχεία μεταξύ, για τις διαφορές μεταξύ των 10 πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, των χωρών μετά τη Μεγάλη Διεύρυνση. Εδώ και πολλά χρόνια ε, αναλύω τις άμεσες ενισχύσεις και ε, ρωτάω τους γεωργούς τι δραστηριότητες δεν θα έκαναν και ε, σε τι αφιερώνουν τις άμεσες ενισχύσεις. Στην Πολωνία τουλάχιστον φαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής των ενισχύσεων αναφέρεται αφορά την τρέχουσα παραγωγή. Πρόκειται για ε, δαπάνες τρέχουσας παραγωγής και 25% μόνο πηγαίνει στις επενδύσεις, στις επενδυτικές δαπάνες και μόνο 5% αφορά δαπάνες που δεν ε, έχουν παραγωγικό χαρακτήρα. Έτσι καταμερίζονται οι άμεσες ενισχύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Πολωνίας. Βλέπετε τα, τη διαφορά στα ποσοστά ανάμεσα στην, στις δαπάνες της τρέχουσης παραγωγής, στις επενδυτικές και στις μη παραγωγικές δαπάνες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στον τρίτο μας καλεσμένο, τον κύριο Ιβ Μάντρα, η Μάδρε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε κυρίες και κύριοι. Μεγάλη τιμή που σας ε, μιλώ. Μιλώ σήμερα λοιπόν ως ε, πρόεδρος της Farmer Αλλά δεν μπορώ να λησμονήσω και την παλαιότερη μου ιδιότητα του Διευθυντή ενό από του κύριου φορεί πληρωμών ενισχύσεων τη κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη. Και άρα έχω και κάποιες ιδέες ε, από αυτή την σκοπιά να σας ε, δώσω. Η οριζόντια ρύθμιση λοιπόν είναι το κλειδί της επιτυχίας της ΚΑΠ που είναι στα χέρια σας ως ε, συνομοθετές και τις επιλογές βέβαια που θα κάνετε ως οι οποίες επιλογές θα ορίσουν αν θα είναι αποτελεσματική, βιώσιμη, διαφανής, διαφανής ως προς τη χρήση του δημόσιου χρήματος ή όλα αυτά σε αρνητικό πρόσημο η κοινή γεωρική πολιτική. Επομένως είναι κατά κύριο λόγο πολιτική επιλογή ε, με την νομοθετική παρέμβαση στην οποία εσείς ε, έχετε τον τελευταίο λόγο. Η πρόταση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας θέτει ενώπιον του εξή διλήμματος. Θα είναι πιο αποτελεσματική η ΚΑΠ για τον Γεωργό, πιο αποδοτική για τον πολίτη πιο αποδοτική για τον φορολογούμενο, πιο αποτελεσματική δηλαδή, πιο ευανάγνωστη, πιο σαφής ως προς τις επιλογές της διάθεσης του δημόσιου χρήματος. Αυτή τη στιγμή η είναι. Είναι ένα σύστημα κανόνων που προσδιορίζονται στις επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τόνισαν νωρίτερα και οι συνομιλητές ε, ως προς τους βασικούς κανόνες αιρεσιμότητας, επιλεξιμότητας, τα μέτρα της ΚΑΠ που προσδιορίζουν και επιλέγουν οι συνομοθέτες και τα οποία μέτρα και κανόνες στη συνέχεια υλοποιούνται ε, μέσα στα κράτη-μέλη από τους γεωργούς και τα επαληθεύουν οι υπηρεσίες ε, καταβολής των ποσών, πληρωμής των ποσών, με τις επαληθεύσεις βεβαίως και των κρατομελών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα έχουμε διπλούς ελέγχους για να επαληθεύεται ότι όλα πάνε καλά και αυτό βέβαια οδηγεί σε αρκετά περίπλοκα συστήματα πολύ συχνά. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα για την μελλοντική ΚΑΠ. Μας λέει ότι θέλει να είναι κάτι πιο ευέλικτο περιστρεφόμενο γύρω από την αποδοτικότητα, το νέο σύστημα, με ένα ευρωπαϊκό σύστημα σαν ε, ομπρέλα, αλλά που επιτρέπει ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν τι εθνικέ στρατηγικές με στόχους εθνικούς, κριτήρια αιρεσιμότητας εθνικά, κανόνες που θα ισχύουν για τα μέτρα όπως αυτά θα έχουν προσδοριστεί από τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, αλλά και πολιτικές ελέγχου κυρώσεων που σημαίνουν πως θα έχουμε 27 διαφορετικά πλαίσια, εθνικά πλαίσια, τα οποία παράγονται από τα κράτη-μέλη, θα επαληθεύονται, θα εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί η Επιτροπή προτείνει να Παρακολουθούνται οι τοποθετήσεις των εθνικών ε, οργανισμών μόνο, ώστε να αποφευθούν οι διπλοί έλεγχοι που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα είναι ένα στοιχείο απλοποίησης για την Επιτροπή αλλά και για τον Γιώργο. Πάντως ο Γιώργος στον καθημερινό του βίο και τη δουλειά θα πρέπει να ε, υφίσταται και τους ελέγχους και τις κυρώσεις ενδεχομένω που θα επιβληθούν και ίσως και περισσότερο από ό,τι τώρα. Γιατί θα καλείται να εφαρμόζει μέτρα, εκτός και αν θεωρηθεί ότι οι εθνικοί οργανισμοί δεν θα κάνουν τίποτα άλλο από το να μετράνε τα εκτάρια στα οποία θα ισχύει το κάθε ε, μέτρο και ότι δεν θα ασχολούνται ούτε με την ορθή καταβολή των ποσών, ούτε με το ενδεχόμενο σφάλμα, ούτε με την επιβολή των ε, συνεπειών ως πρώην διευθυντή οργανισμού πληρωμών, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ή ότι τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια και το ευρωπαϊκό ακόμη θα δέχονταν κάτι τέτοιο χωρί ε, να αντιδράσουν. Ή ότι και ο ή οι συνομοθέτες θα μπορούσαν να δεχθούν ένα τέτοιο ε, διατακτικό, ένα τέτοιο σύστημα στο οποίο θα είναι δυνατόν να επαληθεύεται ότι έχει ορθά δαπανηθεί το χρήμα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου με βάση δηλαδή. Άρα έχουμε ένα άλλο επίπεδο πέραν αυτού του ελέγχου, ένα ετήσιο σύστημα μετρήσεως στατιστικού τύπου, δηλαδή εκτάρια ανά χ ή ύψιλον, ε, ανάλογα με τα μέτρα δηλαδή και το είδος της γεωργικής παραγωγής, που ε, καλείται να τα υλοποιήσει, να υλοποιήσει το κάθε μέτρου, ε, με είτε άρση καθυστέρηση κτλ. τη πληρωμή, σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκληση. Θα υπάρχει και ένα τρίτο σύστημα με βάση δείκτες αποτελεσμάτων που θα έχει πολιτή χαρακτήρα στην επαλήθευσή του. Θα επανέλθω σε αυτό. Και εδώ καλούμεθα να ε, δούμε, να πούμε τι είδου αποτελέσματα παρουσιάζονται με την ε, ΚΑΠ αυτή. Και αν τα αποτελέσματα αυτά τα διάφορα μέτρα και το δημόσιο χρήμα δαπανάται με βάση τους κανόνες και την ε, στόχοθέτηση της ΚΑΠ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο μπορούμε ήδη να συμφωνήσουμε πως υπάρχει ένα θετικό στοιχείο που ενέφερα και νωρίτερα, ότι δεν θα γίνονται διπλή έλεγχη. Αυτό προτείνει η Επιτροπή. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, με λιγότερο σαφείς εγγύησης. Αυτά που συζητεί και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το θέμα της απλοποίησης δηλαδή. Εν τέλει δηλαδή, ο Γεωργός ο οποίος λίγο πολύ θα έχει να υποστεί το ίδιο σύστημα με αυτό που έχει τώρα. Και από την άλλη το κράτος το οποίο θα έχει να κάνει μια επιλογή με κριτήρια αιρεσιμότητας και παρακολούθηση ελπίζω του, οπωσδήποτε της ε, χρηστής του δημόσιου χρήματος αλλά και ένα ε, ε, ετήσιο σύστημα επιδόσεων αυτό το οποίο ανέφερε ο εκδεξιών ε, γειτονά μου που, ως ένα σύστημα με πολύ βαρύ πρόγραμμα παρακολούθησης και επαλήθευση σε ετήσια βάση όπως είπαμε αλλά και εκείνο το πολυετές το οποίο θα έρθει να προσθεθεί στις επαληθεύσεις. Ένα άλλο σημείο με χρήσιμα πιστεύω διδάγματα είναι ότι άπαξ και υπάρχουν 27 όπως ονομάζουμε εθνικοί κανονισμοί με τα κριτήρια της αιρεσιμότητας, της επιλεξιλμότητας και τους ελέγχους και τις κυρώσεις σε εθνικό παντεπίπεδα, υπάρχει κίνδυνο στρέβλωσης από το ένα κράτο στο άλλο και από τον ένα γεωργό στον άλλον. Ενώ τώρα έχουμε μια κοινή βάση. Τελευταίο σχόλιο στη διαφάνεια που βλέπετε έχουν ρόλο να διαδραματίσουν και επιλογές συγκεκριμένε στο τωρινό σύστημα οι συνομοθέτες και με το καινούριο σύστημα εσείς συνομοθέτες κοινοβούλιο και συμβούλιο παραμένετε μόνο ως λογιστική απογραφής της αποτελεσματικότητας μεγαλύτερη σημεία του νέου συστήματος σε σχέση με τους γεωργούς που το εκτελούν. Η ΚΑΠ λοιπόν με τη στοχοθέτηση των επιδόσεων και την υπόσχεση προς τον πολίτη ότι θα μετράμε την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητά της και θα αποδεικνύουμε τη χρησιμότητα της κάθε δαπάνης σε ευρώ που έχει εγκριθεί. Αυτή λοιπόν η νέα ΚΑΠ τι σημαίνει τελικά ότι θα γίνεται μια ετήσια στάχδη μέτρηση της αποδοτικότητας, δηλαδή σε όρους στατιστικούς και μόνο, με ένα πολιετές επιπλέον σύστημα, το οποίο θα συνδέεται με ένα σύστημα δικτών αποτελέσματος και για να ε, χρησιμοποιήσω και το κείμενο της πρότασης, δείκτες αποτελέσματος οι οποίοι δεν βλέπω να επιτρέπουν την ε, προσμέτρηση αποτελεσμάτων. Και αυτό που με προβληματίζει και πιστεύω θα πρέπει να είναι και δικό σας προβληματισμός ή πρόβλημα και για σας. Τι θα συμβεί, ε, ένα διατακτικό που θα πρέπει να αξιολογηθεί σε διάμεση φάση, πώς θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για την οικονομική και περιβαλλοντική αποδοτικότητα της νέας ΚΑΠ. Δηλαδή θα λέμε σε τόσα εκτάρια, στην περιοχή α, β, γ, με τους γεωργούς που ακολουθούν το α ή το β ε, σύστημα ή σύστημα μέτρων, πώς θα μπορούμε να πούμε ότι αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ε, ελπίδες που έχουν γεννηθεί σε σχέση με την αποδοτικότητα αυτού του συστήματος. Χρειάζεται πραγματική δουλειά να έχουμε δείκτες, λίγους μεν, αλλά δείκτες γνήσιας απόδοσης και αντικτύπου. Δείκτες αντικτύπου που θα προσμετρούν την απόδοση και αποδοτικότητα της ΚΑΠ στο μέλλον μέσα σε μία γενική πολιτική που θα κάνει μέτρηση πολύ πολυετή και εδώ ακριβώς βλέπουμε ότι ε, έγκυται, και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και για να ολοκληρώσω κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, το διτακτικό αυτή τη στιγμή βλέπω να έχει δύο θετικά στοιχεία. Το στοιχείο δηλαδή της εθνικής στρατηγικής που λέει ότι τα κράτη-μέλη καλούνται να κάνουν ε, επιλογές πολύ πιο συνεκτικές μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Και δεύτερο θετικό στοιχείο, ότι έχουμε πιο συγκεκριμένη μέτρηση από την ΚΑΠ του αντικτύπου των μέτρων που αυτή ε, χρηματοδοτεί. Στο πλαίσιο αυτό όμως, μένει πάρα πολύ δουλειά να γίνει για να προσδοριστούν οι δείκτες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αρκεστούμε στους δείκτες όπως αυτοί τώρα προτείνονται που είναι δείκτες αποτελέσματος, όχι γνήσιοι όμως, όχι αυτό που θα εννοούσαμε με τον κοινό όρο δείκτες αποτελέσματος. Με ένα διατακτικό το οποίο θα έπρεπε ε, να μας οδηγεί ως ε, φορολογουμένους να απαιτούμε χρηστή δαπάνη των δημοσίου χρήματος, αλλά και ταυτόχρονα την ανάγκη για τους γεωργούς της Ευρώπης να έχουν μια πιο γερή βάση και ενιαία βάση πολιτικής για τη γεωργία. Και σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από, για τη λύση στο πρόβλημα αυτό, από κανόνες πιο απλούς, κανόνες που θα προσδορίσουν οι συνομοθέτες και αντιλαμβάνουμε ότι αυτή είναι η δική σας προσπάθεια μέσα από τους αφορούς κανονισμούς, με κανόνες απλούς όπως είπα, που θα προσδορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο, με στοιχεία που θα προσδορίσουν τι είδους έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται στα κράτη-μέλη με κοινή βάση και με κυρώσει κοινέ. Δεν θα ακολουθείτε δηλαδή μεταβλητή γεωμετρία από το ένα κράτος μέλο στο άλλο. Γιατί πρέπει με αυτό το βασικό κόρπου κανόνων, είτε είναι η επιλεξιμότητα, η αρισμότητα για τους γεωργούς, ε, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορούν να διαφοροποιούν τα κρατημέλη. Πρέπει να ε, έχουμε μέτρα λίγο πολύ κοινά και με αποτέλεσμα λίγο πολύ ισοδύναμο από το ένα κράτος στο άλλο. Και αυτό νομίζω δίνει ταυτόχρονα απαντήσεις και στην ανάγκη για ευελιξία. Η πρόταση της Επιτροπής, η πρόταση Επιτροπής που έχει να κάνει με τον έλεγχο για, τις, ε, για τους φορείς πιστοποίησης είναι ένα στοιχείο απλούστευσης, πρέπει να υποστηριχθεί και εάν τυχόν ε, μπορώ να προλάβω το ερώτημα, γιατί να μην γίνεται με την τωρινή ΠΑΚ. Μα θα μπορούσε. Θα μπορούσε και αυτό θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην απλοποίηση και για την τωρινή ΠΑΚ. Και αν μιλούμε για μια ΚΑΠ ε, αποτελεσμάτων και επιδόσεων, πρέπει να περάσουμε σε μια πολυετή αξιολόγηση, γιατί η ενιάμψη αξιολόγηση δεν, δεν επιτρέπει ε, ανάγνωση σωστή των αποτελεσμάτων. Πρέπει να έχουμε πολυετή αξιολόγηση, με δείκτες όμως λογικούς, σωστούς, που θα, θα αποδεικνύουν και το οικονομικό αλλά και το περιβαλλοντικό όφελος από τα μέτρα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ασφαλώς, ε, πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων μπροστά μας, αλλά πρέπει οπωσδήποτε, και μιλήσατε νωρίτερα και για τα, η ψηφιακή τεχνολογία στο προηγούμενο κομμάτι της συνεδρίας Δεν είμαστε σε μια Ευρώπη όπου, έχουν, όπου θα έχουν περάσει στο 100% της ψηφιοποίησης όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό, αυτό υπολοιπόμεθα. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε πρόσθετα ο δίκτυ να φανταστούμε μια μέση αξιολόγηση της μετάβασης στη νέα τεχνολογία. Να πούμε, δηλαδή έχουμε τόσες ε, εκμεταλλεύσεις ή τόσους γεωργούς που περνούν στη νέα τεχνολογία. Ας υπάρχει όμως, για όνομα του Θεού, ένας δείκτης επιδόσεων που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών και που θα είναι συνεκτικός με την ίδια βάση για όλους για να έχουμε ένα σύστημα ισορροπημένο, μία ΚΑΠ ισορροπημένη χρειάζεται ένα σύστημα πολυετές που θα, υπο, θα υπολογίζει, θα καταγράφει, θα κάνει απολογισμό των επιδόσεων της ΚΑΠ και αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ και περνάμε στη συζήτηση, στις ερωτήσεις ε, των Ευρωβουλευτών. Παρακαλώ δηλώστε αν θέλετε το λόγο. Φλάναγκαν για να δούμε πόσο, πώς θα κατανείμουμε το χρόνο. Να γνωρίζουμε πόσοι θέλουν το λόγο. Άγνιου Γιάρ. Άγνιου Καϊ. Χουμόκ. Παμ Νταμτέ. Νταμτά. Άγνιου, Ντεκάστρο, Φλάναγκαν, Γιάρ και χουμοκ παμ νταμτε Νταντά. αγνιου φλαναγκαν γιαρ κανείς? Αντριέ. Ωραία. Έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε τρία λεπτά το πόλιο ο καθένας παρακαλώ. Ο κύριος Άγνιο. Τρία λεπτά κύριε Άγνιο. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κάποιες ερωτήσεις προς τον δεύτερο ομιλητή και μία προς τον τρίτο. Ο δεύτερος ομιλητής από την Πολωνία έρχεται και μίλησε για το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μία από τις κατηγορίες ήταν η μικρή εκμετάλλευση, όπου ε, το εισόδημα του γεωργού είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο εισόδημα οι εκμεταλλεύσεις ε, στην Πολωνία που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία ε, είναι όπως στη Γαλλία και τη Γερμανία όπου αυτός που μένει εκεί εργάζεται σε κάποιο εργοστάσιο για παράδειγμα και απλά έχει την εκμετάλλευση ως χόμπι λίγο πολύ, ως ασχολία του Σαββατοκύριακου. Ε, και η δεύτερη ερώτηση προς εσάς είναι υπάρχει ο πυλώνας 2, ε, τα περιβαλλοντικά προγράμματα και στη Βρετανία. Πολλοί γεωργοί αποθαρρύνονται από τα προγράμματα αυτά λόγω της πολλοπλικότητάς τους. Ε, και εγώ ίδιος έχω δαπανίσει πολλά χρήματα ε, για τα προγράμματα αυτά χωρίς να μου έχει επιστραφεί ούτε δραχμή, <laughs> που λέει ο λόγος. Και η ερώτησή μου προς τον τρίτο ομιλητή είναι το θέμα των ε, πληρωμών, των ενισχύσεων με βάση ε, τις επιδόσεις. Έχουμε αναθέσει στους ε, γεωργούς να μετριάσουν την αλλαγή του κλίματος, δηλαδή να καλλιεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί το κλίμα. Πώς μπορούμε να περιμένουμε από ένα γεωργό να αποδείξει ότι ο τρόπος που καλλιεργεί τα προϊόντα του βελτιώνουν τον καιρό. Νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό αυτό και ελπίζω έτσι να δείξουμε πόσο μεγάλη ανοησία είναι όλα αυτά. Κύριε Στεκάστρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους τρεις καλεσμένους, τους τρεις εμπειρογνώμονές μας, γιατί μας έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Έχω μία ερώτηση προς τον τρίτο καλεσμένο μας, τον κύριο Ιβ Μάντχα αν κατάλαβα καλά, η πρόταση του οριζόντιου κανονισμού αφήνει τη διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη για να προβλέψουν τους στόχους τους και να δουν με τι μέσα θα υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους και επίσης να αξιολογήσουν αν τα μέσα ε, ήταν ικανά για την υλοποίηση των στόχων. Και όλα αυτά στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους. Αν τώρα κατάλαβα καλά και αν αυτή όντως είναι η προσέγγιση, τι κίνδυνο διατρέχουν τα κράτη-μέλη. Κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων. Ε, και τι θα γίνει αν ε, καταλήξω συμπέρασμα ότι δεν υλοποιήθηκε ο στόχος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν κάποιες οικονομικές διορθώσεις. Και στη συνέχεια, αν αυτή όντω είναι η προσέγγιση, τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη που έχουν περιφερειακή οργάνωση, που συνταγματικά δηλαδή προβλέπονται περιφερειακές αρμοδιότητες. Οπότε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους της, τα μέσα της και να καθορίσει ε, ποια εταιρεία θα κάνει την αξιολόγηση της υλοποίησης αυτών των στόχων, ποια πιστοποιημένη εταιρεία θα κάνει ε, την αξιολόγηση. Και αν όλα είναι έτσι όντως, τότε τι απλούστευση μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το σύστημα. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ πολύ για και τις τρεις παρουσιάσεις. Κρίμα που δεν ήταν εδώ παρόντες περισσότεροι, διότι πολλά είχαμε να μάθουμε από αυτές τις παρουσιάσεις. Ε, πάντως, εγώ όπως αντιλαμβάνομαι ε, το ότι κάτι στηρίζεται σε επιδόσεις είναι ότι λαμβάνει κανείς ε, χρήματα ανάλογα με τις επιδόσεις του. Νομίζω ότι είναι δίκαιο το σύστημα. Νομίζω ότι έτσι παρακινεί τους ανθρώπους να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και και όσοι καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες ανταμείβονται γι' αυτό. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για σύγκληση δεδομένου ότι το, η πρόταση αυτή λέει ότι μέχρι το τέλος τη επόμενη ΚΑΠ θα έχουμε ε, συμμόρφωση κατά 75% ε, ε, γιατί να λαμβάνουν κάποιοι το 75% και άλλοι το 100% εάν ε, και, ο μεν, και οι μεν και οι δε έχουν εξίσου καλές επιδόσεις. Ευχαριστώ. Äh, ο κύριο Σιγιάρ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ για χρονικού λόγου μπόρεσα να παρακολουθήσω μόνο την τελευταία ομιλία. Ερώτηση όμω προ και του τρει ομιλητέ. Υποθέτω ότι συμφωνούμε και ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα οδηγήσει σε μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, το σύστημα αυτό όμως ε, ενέχει μεγάλους κινδύνους. Έχουμε μια ελπίδα απλούστευσης της γεωργίας με το σύστημα αυτό και εάν ναι πώς. Εάν δεν έχουμε απλούστευση τότε δεν έχουμε και κανένα όφελος. Δεύτερη ερώτηση, περιγράψατε τους κινδύνους. Έχουμε κοινού στόχους, έχουμε κοινού δείχτες, έχουμε ένα κοινό σύστημα. Τα κράτη-μέλη ήδη εκπονούν ε, εθνικά στρατηγικά σχέδια. Όλα αυτά πώς συνδυάζονται στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής, ώστε να μην έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα Είπατε ότι καταρχά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν αποτελέσματα στην Κομισιόν, ε, θα πρέπει να υποβάλουν ε, ε, τα σχέδιά τους και κατόπιν να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εγώ προσωπικά φοβάμαι, εάν έχουμε εθνικά στρατηγικά σχέδια, η Γερμανία να σας βάλει ένα έγγραφο που να ζυγίζει 10.000 κιλά, ενώ άλλοι να σας δώσουν ένα δεκασέλιδο έγγραφο. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιον βαθμό εναρμόνισης στο θέμα αυτό. Τρίτη ερώτηση. Ε, έχουμε από τη μία ε, αναθεώρηση της σχέσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Και έτσι έχουμε το πλαίσιο επιδόσεων με δείχτες. Ε, και από την άλλη έχουμε τη σχέση ανάμεσα στο κράτος μέλος και τους γεωργούς. Πώς μπορούμε να απλουστεύσουμε την ε, σχέση αυτή ανάμεσα στον οργανισμό πληρωμών και τον γεωργό. Έχετε κάποια πρόταση. Και φοβάμαι όσον αφορά τους στόχους ότι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον στόχο αναγεωργό, αναγεωργική εκμετάλλευση. Πώς λοιπόν θα λειτουργήσει το κράτος μέλος ως ε, ε, μεσολαβητής. Δεν είναι απόλυτα σαφές αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε τον αριθμό των σελίδων των σχεδίων των διαφόρων χωρών. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ο κύριος Δάντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ ε, και τους τρεις ομιλητές σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Έχουμε να απαντήσουμε στα εξή στα ερωτήματα με βάση τρία σημεία εισόδου. Καταρχάς, τη συνθήκη που στηρίζει τη συνθήκη της Ρώμης ε, και που δίνει μια ιδιαίτερη φρομέριμνα για τη γεωργία, παραγωγή προϊόντων ποιοτικών για τον καταναλωτή και σε τιμές οικονομικά άνεκτες. Μας έχουμε ένα πρώτο οικονομικό στοιχείο. Δεύτερον, η ΚΑΠ αμφισβητείται αυτή τη στιγμή από ένα τμήμα της ε, κοινή γνώμης που θεωρεί ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα φιλοδόρημα ή με ένα μπαξίσι προς τον ε, Γεωργό, εφόσον είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ευρωπαϊκού Προπολογισμού η ΚΑΠ, επομένω, χρειάζεται αυτή η οικονομική σχέση να είναι και προσεκτική. Επομένω, ρωτώ και του τρεις ομιλητές ε, τι θεωρούν ότι μπορεί στην προσεχή προγραμματική περίοδο να συμβεί εάν δεν προκύψει μια πραγματική έγκριση των λογαριασμών επειδή θα υπάρχουν ε, δείκτες ε, δημοσιονομικοί από το ελεγκτικό συνέδριο. Και τρίτον, βλέπουμε να συμβαίνουν ανά τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη, εξελίξεις κλιματικές που είναι καθημερινές και που μας προβληματίζουν και ταυτόχρονα και με την εξέλιξη της βιοποικιλότητας πρέπει η Γεωργία μέσω των πολιτικών της να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα νέα ε, σε αυτούς τους νέους προβληματικούς και τα νέα αυτά διακυβεύματα θεωρείτε ότι αρκεί όλο αυτό το πλαίσιο για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννώνται και για την κοινωνία με την κλιματική αλλαγή αλλά και σε σχέση με, τους λοιπούς, με τα λοιπά ζητήματα και τι προτάσεις θα μπορούσατε να μας κάνετε για τα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Κύριος Αντριού, ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους, ε, τέσσερις, τους τρεις ομιλητές μας βλέπουμε την έννοια της απλοποίησης και της επικουρικότητας να ε, επιλέγονται ε, ως ε, καθοριστικοί παράγοντες, αλλά αυτά που μας είπατε δεν με, καθορι... δεν με τους προς τον άλλο παράγοντα. Έτσι λοιπόν διερωτώ με, χρειάζεται επιτακτικά να επανεθνικοποιηθεί, γιατί ως περί αυτού ουσιαστικά πρόκειται η γεωργική πολιτική, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μέσα από μια πραγματική κακινή πολιτική τον δείκτη της, ε, των επιδόσεων στο βάθρο αυτής της πραγματικά κοινή και κοινοτική πολιτικής. Ή να το πω αλλιώ, τι, ε, τι το καινούριο θα έμενε ε, σε σχέση με αυτή την μεταρρύθμιση που μας παρουσιάζεται σήμερα. Ένα άλλο σημείο, η δυνατότητα και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντοντέν, ε, η δυνατότητα λοιπόν να δοθούν απαντήσεις και δεδομένων και των κλιματικών αλλαγών σε, όλα, ε, σε όλες τις προκλήσεις που είναι εξωτερικές της ε, κοινωτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε σε οικουμενικό επίπεδο στοιχεία που μπορεί να μας οδηγήσουν σε περισσότερη φτώχεια εδώ τους Ευρωπαίους γεωργούς. Και επομένως, και τρίτο ερώτημα, πώς μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη αυτή η μεταρρύθμιση όπως παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Δύσκολα τα πράγματα αυτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, ο κύριος Μαγκέρερ. Ο Μέγκελε, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω μέσα σε λίγα λεπτά να συνοψίσω τις απαντήσεις που πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσω στις παρουσιάσεις και να απαντήσω και σε μια σειρά ε, ερωτήσεων που τέθηκαν. Να ξεκινήσω πρώτα από μία δήλωση του φίλου μου, του Ιβ Μάντρε, που είπε ότι θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που να, ε, που να εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες σε, σε όλους. Νομίζω ότι αυτό ήδη είναι περιγραφή της ε, πολιτικής ε, όπως ε, ισχύει σήμερα. Δεν μιλώ για το δεύτερο πυλώνα, διότι ο δεύτερος πυλώνας είναι πολύ διαφοροποιημένος. Γι' αυτό άλλωστε έχει φτιαχτεί. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη ε, να ε, προσαρμόζουν ε, τους κανόνες, αλλά υπάρχουν 40 ή 50 διαφορετικοί τρόποι να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη τον πρώτο πυλώνα της άμεσης ενισχύσης. Και αν συγκρίνει κανείς το σύστημα άμεσων ενισχύσεων στη Γαλλία με αυτό στη Γερμανία, δεν θα βρει πολλέ ομοιότητε. Ε, ισχύει λοιπόν και δεν ισχύει ότι ε, οι ίδιοι κανόνε ισχύουν για όλους. Δεύτερον, ε, η απλούστευση έχει αμφισβητηθεί, δεν υπάρχει εγγύηση απλούστευσης. Γιατί είναι τόσο πολύπλοκη η πολιτική σήμερα. Διότι βασίζεται αποκλειστικά σε κανόνες και ο η εφαρμογή των κανόνων ελέγχεται προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζεται ένας μηχανισμός ε, εκπόνησης όλο και πιο αναλυτικών κανόνων και αύξησης των ελέγχων κάθε φορά που εντοπίζονται λάθη και παραλήψεις. Και μιλώ από προσωπική πείρα, διότι τα τελευταία 8 χρόνια είμαι αρμόδιος για το τμήμα ελέγχου. Και έτσι Τελικά ο Γεωργός υφίσταται όλη την αυστηρότητα του νόμου και κανένας ε, δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό διότι κάθε επίπεδο του συστήματος αυτού παραπέμπει στο ανώτερο επίπεδο και λέει ότι ε, αν δεν το κάνω αυτό θα με τιμωρήσει ο ανώτερο. Και συχνά λέμε το ίδιο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εδώ στο Κοινοβούλιο ε, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θέλουμε να ε, σταματήσουμε αυτή την πρακτική. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε απλούστευση εάν δεν ξεφύγουμε από τον τεράστιο αριθμό κανόνων που εφαρμόζεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Η άλλη μου παρατήρηση έχει να κάνει επίσης με μια δήλωση του Ιβ Μάντρε, γιατί δεν εφαρμόζουμε ήδη τους οργανισμούς πιστοποίησης ε, και, τον, ε, και την ενιαία προσέγγιση ελέγχου. Μα το κάνουμε αυτό. Το 2015 ξεκινήσαμε και έκτοτε... Οι έλεγχοι μας βασίζονται όλο και περισσότερο στα αποτελέσματα των οργανισμών πιστοποίησης, αλλά χρειάζεται χρόνο ένα τέτοιο σύστημα, διότι πρέπει να ελέγχει την ποιότητα δουλειάς των οργανισμών πιστοποίησης. Εάν μεταφέρουμε αυτό το σύστημα στο νέο μοντέλο υλοποίηση θα μπορέσουμε να βασιζόμαστε όλο και περισσότερο στις εργασίες των οργανισμών, πληρωμών, ε, οργανισμών πιστοποίησης από ό,τι σήμερα σε όλες τις παρουσιάσεις αλλά και σε όλες τις ερωτήσεις λείπει ένα στοιχείο που είναι στοιχείο κλειδί για τη μεταρρύθμιση που είναι η έγκριση των σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ακούγοντας ε, σήμερα τις παρεμβάσεις ε, στη συζήτηση ότι τα κράτη-μέλη συντάσσουν το σχέδιό τους ε, και τελείωσε. Όχι, αντιθέτως πρέπει τα κράτη-μέλη να περάσουν από ανάλυση των αναγκών τους και αυτή είναι μια διαδικασία που συνοδεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποβάλλουν τα σχέδια τους, ε, ε, τα οποία συζητώνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό έχει θεσπίσει μια σειρά κριτηρίων για επαλήθευση και ελέγχου που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πούν στα κράτη-μέλη ότι στο τάδε και το τάδε σημείο δεν συμμορφώνονται όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ε, την απλούστευση του συστήματο. κλπ. Δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια αυτά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ε, όσον αφορά τη συνολική πολιτική. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη έχουν πάρα πολλέ επιλογέ που μπορούν να εφαρμόζουν αυτόνομα. Στο μέλλον θα έχουμε επιλογέ που θα μπορούν να εφαρμόζουν στο πλαίσιο ε, μια διαδικασία προγραμματισμού που τελειώνει με την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι θα έχουμε περισσότερα κοινά στοιχεία από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή στην κοινή γεωργική πολιτική όπω εφαρμόζεται σήμερα. Η επόμενη μου παρατήρηση είναι ότι λείπει συστηματικά εδώ ένα στοιχείο κλειδί που είναι η ερώτηση θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε εάν τα κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν ε, τους ε, κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις βασικές απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ναι, αυτό γίνεται με συστηματικούς ελέγχους και εάν διαπιστώσουμε ότι το κράτος μέλος έχει ένα σύστημα ελέγχου το οποίο δεν συμμερφώνεται με τους κανόνες αυτούς, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές δράσεις. Αυτό είναι απαραίτητο για να φροντίσουμε να παραμένουμε η πολιτική αυτή κοινή. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο νομιμότητας, ε, όχι όμως πια σε επίπεδο ε, ε, επιμέρους δικαιούχων και το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να σπάσουμε το φαύλο κύκλο, να έχουμε όλο και πιο πολύπλοκους κανόνες ε, που να καταλήγουν σε επίπεδο δικαιούχου, αλλά ε, να έχουν να κάνουν με τη σχέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, έχουν υποβάλει την γνωμοδότηση, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της νομοποίησης, ε, της ενών, της, ε, της νομιμοποίησης και θα ήθελα να πω ότι νομοθέτης δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το ελεγκτικό συνέδριο. Ο νομοθέτης θεσπίζει τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα όσον αφορά την ενίσχυση, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και εμείς έχουμε συντάξει τις προτάσεις μας με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν τις ε, εγκρίνεται να υπάρχουν σαφείς κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αλλιώς απλά αφήνεστε στα χέρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα καθορίσει μεγάλο τμήμα της πολιτικής αντί να το κάνει αυτό ο νομοθέτης που είναι αρμόδιος θα δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου τον κύριο Λοντέρο που θα μιλήσει για τις πτυχές που συνδέονται με τις επιδόσεις στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να προσθέσω κι εγώ κάνα δύο σημεία για το νέο πλαίσιο των επιδόσεων και το, την ομάδα δικτών που προτείναμε για να καταμετρούμε σε κάθε φάση της επιδόσεις. Καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι δεν επανεφίβραμε τον τροχό. Το σύστημα αυτό υπάρχει ήδη. Και σε αρχές του Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ε, μια πλήρη δεσμή δεδομένων για τους δείκτες ε, του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Και είναι τα αυτά τα στοιχεία, όλοι οι δέσμοι, αλλά έχουμε και διαδραστικά dashboards που βλέπετε ε, ποια είναι τα αποτελέσματα των διαφόρων επεμβάσεων. Και με την έκθεσή μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση της ΚΑΠ ε, με το τρέχον σύστημα. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω μια βασική αλλαγή στην πρότασή μας. Τα εθνικά σχέδια για την κοινή πολιτική θα πρέπει να εξετάζονται από το πρίσμα των στόχων, όχι των μέσων. Ε, δηλαδή, τις επιδόσεις πολιτικής τις, τις κρίνουμε με βάση τους κοινού μας στόχους και όχι τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων. Οπότε, οι κανόνες προβλέπουν μια κοινή δέσμη στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα ιδιαίτερες ανάγκες στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες, και υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τον, εντο, για τον εντοπισμό για την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων με βάση τις ιδιαιτερότητες και γι' αυτό μπορεί κανείς να επιλέξει την α ή β παρέμβαση. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων από δύο ταμεία, από δύο γεωργικά ταμεία, οπότε είναι πολύ πιο ευρύ το περιθώριο των παρεμβάσεων. Η εμβέλεια των παρεμβάσεων είναι ευρύτερη. Επίσης, ε, υπάρχει μια συνοχή στη νέα προσέγγιση που δεν είναι δεδομένη βέβαια, θα συζητηθεί στη συνέχεια και θα αξιολογηθεί. Αυτή είναι μια κρίσιμη φάση της διαδικασίας η αξιολόγηση. Και κατόπιν, σε αιτήσια βάση, έχουμε συστήματα υποβολής εκθέσεων που δίνουν την παραγωγή, ε, τη χρησιμοποιούμενη έκταση, το ύψος των άμεσων ενισχύσεων, τους δικαιούχους, ε, το ύψος των δαπανών. Και έχουμε και δείκτες αποτελεσμάτων. Ε, γιατί κάθε παρέμβαση έχει ένα σκοπό. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να κριθεί με βάση τα αποτελέσματα η κάθε παρέμβαση. Ξέρουμε ότι μία παρέμβαση είναι υποφελής για τη βιοπικιλότητα. Οπότε μπορεί ένα κράτος να θέλει να αυξήσει τον αριθμό των εκταρίων που υπάγονται σε αυτή την πρακτική. Και υπάρχει και ένα τρίτο στρώμα, ε, οι δείκτες αντικτύπου, οι δείκτες επιπτώσεων, που καταμετρούν τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της πολιτικής. Και αυτό είναι πιο δύσκολο βέβαια να καταμετρηθεί. Όλοι συμφωνούμε. Γιατί όταν το αποτέλεσμα είναι πολύ και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ε, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ποιο είναι ποιε είναι οι επιπτώσει τη κάπη των άλλων παραγόντων. Πάντω, το πλαίσιο των επιδόσεων, το νέο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα μα επιτρέψουν να κρίνουμε κατά τη στιγμή έγκριση του σχεδίου, αν είναι το σχέδιο αυτό φιλόδοξο, αν είναι σωστό για τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχει το κράτο μέλο και υπό το φω τη υλοποίηση των κοινών μα στόχων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Μετά τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δημιουργήθηκαν ε, νέες απορίες. Για να σας δώσω από ένα λεπτό στον καθένα να τις υποβάλλετε αν θέλετε. Ο κύριος Γιάννης ζήτησε το λόγο, αλλά ένα λεπτό παρακαλώ αυστηρά. Ναι, θέλω απλώς να υποστηρίξω το γεγονός ότι όλοι νομίζω έχουμε σαν μέλημα το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως τα κράτη-μέλη αφού θα έχουν διατυπώσει τις εθνικές στρατηγικές θα μπορούν να επιτρέψουν την ύπαρξη ακόμη μιας κοινή γεωργικής πολιτικής. Το είπατε κι εσείς μόλις τώρα ότι πρέπει να προσέξουμε αυτή η κοινή γεωργική πολιτική να μην ε, κατακαιρματιστεί σε 27 διαφορετικές εθνικές γεωργικές πολιτικές. Έχουμε υποτίθεται ένα κοινό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, την κοινή γεωργική πολιτική. Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να ανησυχούμε εδώ στην Επιτροπή ότι μπορεί να μας ξεφύγει ο έλεγχος αυτού του πλαισίου από τα χέρια μας. Ναι, αλλά πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε κάποια ευελιξία. Και μέχρι στιγμής κατηγορούσαμε την προηγούμενη πρόταση για έλλειψη ευελιξίας, για ανελαστικότητα και για μικρή επιρροή του κράτους γιατί όλα περνάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εγκρίνει τα στρατηγικά σχέδια. Και αν διαπιστώσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή της ανταγωνιστικότητας, τότε ε, θα ξεκινήσει συζήτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συγκεκριμένου κράτους, το σχέδιο του οποίου έχει διατυπωθεί, έχει εντοπιστεί ένα πρόβλημα. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που μας είπε ο κύριος Μέγκελε. Και θα ήθελα να τον καθησυχάσω σε ό,τι αφορά την ερώτησή μου για το ελεκτικό συνέδριο. Ξέρετε κύριε Μόγγελε ότι ε, όταν το ελεκτικό συνέδριο προσπαθεί να σφετεριστεί το έργο μας, ε, μας ε, εκνευρίζει ιδιαίτερος. Και φαντάζομαι αντίστοιχο φόβο έχει και το ελεκτικό συνέδριο. Θα κάποιο φετερίσει το δικό του έργο. Και πολλά τα μάλλον που βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και μερικέ φορές υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών που ακούμε επί τόπου και αυτών που ακούμε, αυτών που ακούμε εδώ. Γιατί το θέμα των κοινοτικών κονδυλίων και πώ χρησιμοποιούνται δεν είναι ένα ερώτημα που αφορά μόνο το ελεγκτικό συνέδριο. Και εμείς θα πρέπει να δούμε αν πιάνουν τόπο τα χρήματα και πού πηγαίνουν. Και μάλιστα η υπηρεσία Σολάφ εντόπισε ένα πρόβλημα στην Κορσική για καμιά δεκαετία παραγωγούς. Νομίζετε ότι κάποιος δεν θα μας το ρωτήσει αυτό ε, στην προεκλογική εκστρατεία, δεν θα μας ρωτήσει γιατί δεν γίνονται περισσότεροι έλεγχοι στις πληρωμές και ποιος κάνει αυτούς τους ελέγχους. Πώς λοιπόν θα βεβαιωθούμε ότι γίνεται η ίδια χρήση των κονδύλιων στα κράτη-μέλη και θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι πιάνουν το από παντού τα χρήματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όποιος δεν ενδιαφέρεται πήρε τα χρήματα από τη συμμόρφωση. Το θέμα είναι σε ποιον δίνονται τα χρήματα, ποιο είναι ο δικαιούχο των κονδύλιων, πώ πανονται τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ανδρία. Ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι μόνο μετά τις ομιλίες που ακούσαμε. Μπορείτε να μας πείτε σε που έγκυται η απλούστευση της μεταρρύθμισης της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής για το Γεωργό. Εντάξει, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβα τι απλούστευση υπάρχει και πώς την εξυπηρετεί, αλλά για το δικαιούχο το Γεωργό δεν βλέπω που έγκυται αυτή η απλοποίηση. Πώς θα τη νιώσει την απλούστευση ο Γεωργός στο χωράφι του με την νέα μεταρρύθμιση κάπου. Ο κύριος Φλάναγκα. Εξαιρετική ερώτηση και θέλω πάρα πολύ να ακούσω την απάντηση. Και η ερώτηση που έθεσα ε, στους ομιλητές ήταν η εξή και ίσως η Κομισιόν μπορεί να μου απαντήσει. Αν έχουμε ένα σύστημα που να βασίζεται στις επιδόσεις, μπορεί κανείς να μου εξηγήσει τη λογική της σύγκλησης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς ε, στο τέλος αυτής της, κοινής, αυτής της περίοδου ε, θα λαμβάνει κάποιο μόνο το 75% σε σχέση με κάποιον άλλον με τις ίδιες επιδόσεις. Πώς μπορεί αυτό να βασίζεται στις επιδόσεις. Η και εγώ έχω μια ερώτηση. Με τους κοινού κανόνες θα πρέπει να δημιουργούμε παρόμοιες ευκαιρίες, δυνατότητες και ωφέλη για τόσο διαφοροποιημένη γεωργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί οι κοινοί κανόνες, οι ενιαίοι κανόνες για τόσο διαφορετικά μοντέλα γεωργίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου είναι εφικτό. Είναι δυνατό λοιπόν να έχουμε κοινούς κανόνες που θα ισχύουν σε τόσο διαφοροποιημένα είδη γεωργίας, άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και με τόσο διαφορετικές περιστάσεις στη γεωργία. Πέντε λεπτά λοιπόν θα δώσω στους καλεσμένους και στους προσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λιγότερο μπορείτε, περισσότερο δεν γίνεται. Θα ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτο ή από τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες. Ίσως αυτή τη φορά καλύτερα να ξεκινήσουμε από τους εμπειρογνώμονες μας. Ξεκινάμε από τους εμπειρογνώμονες, λοιπόν. Με ποια σειρά θέλετε να μιλήσετε. Ο κύριος Μάντρα. Σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας πρώτη είναι καλύτερη πάντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κάποιο πρέπει να κάνει την αρχή, λοιπόν. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις απαντήσεις στα διάφορα κεφάλαια που έχουν διατυπωθεί. Επανεθνικοποίηση και εναρμόνιση, αν μπορεί να υπάρχουν κοινέ διατάξεις, με σεβασμό όμως και των διαφορετικών πλαισίων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε και να επαναλάβουμε πως η ΚΑΠ με τον πρώτο πυλώνα είναι κατεξοχήν κοινοτική. Εδώ υπάρχει ένα σαφές σημείο απόκλησης. Ο βασικός καρόνας της αιρεσιμότητας και του πρασινίσματος και το 60% των βοήθητων ενισχύσεων με τον πρώτο πυλώνα δεν ανήκουν στα κράτη-μέλη, δεν είναι στα χέρια των κρατών μελών. Αυτό ορίζουν οι κανόνες που έχουν επιβάλει οι συνομοθέτες. 5% του πρώτου πυλώνα με την ευελιξία που έχει χορηγηθεί ανήκει στα κράτη-μέλη. Με την πρόταση λοιπόν που γίνεται εδώ, η ευελιξία από το 37% πάει στο 98%. Άρα αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Επίσης μπορούμε να έχουμε κάτι το κοινό δίνοντας ταυτόχρονα απάντηση στις ιδιαιτερότητες για το Γεωργό ή για την ε, Ήπεθρο που είναι πολύ διαφορετικές, στις πραγματικότητες που είναι πολύ διαφορετικές. Ναι, μπορούμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, δηλαδή μια κοινή απέτηση βάσεως. Τι απαιτεί η ΚΑΠ από τον κάθε Γεωργό, τι πρέπει να κάνει κατελάχιστον, τι πράγματα πρέπει να σέβεται κατελάχιστον. Εάν όμως επιβάλλουμε αυτήν την κοινή απέτηση ως βάση, μπορούμε ταυτόχρονα να θέσουμε και ένα διατακτικό ισοτιμίας που θα αξιολογεί αυτή την αποτελεσματικότητα. Αλλά μόνο εάν ξέρουμε η ισοτιμία μας σε τι αντιστοιχεί. Ιδάλλως, αν δεν το ορίσει αυτός ο νομοθέτης, ισοτιμία σημαίνει τα πάντα ή τίποτα. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια επιλογή. Επίσης λέγεται, και εδώ πάλι έχουμε μια πρόταση, ένα στοιχείο της πρότασης δηλαδή, ότι θα έχουμε 27 τουλάχιστον εθνικά στρατηγικά σχέδια, 27 εθνικές γεωργικές πολιτικές. Αλλά, αλλά μας λέτε, μας λέγεται, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που πρέπει να γίνεται σεβασμό κατά κύριο λόγο και καταρχήν από την έγκριση της Επιτροπής που επαληθεύει τον κοινό στόχο πολιτικής. Μάλιστα. Αλλά όταν έχουμε μια σαν κυβέρνηση, ισχύρη κυβέρνηση, με ιδιαίτερες δυσκολίες και με ευαισθησίες διακυβέρνησης περισσότερο ή λιγότερο υψηλέ ή έντονε σε σχέση με το περιβάλλον και την οικονομία κτλ. Θα είναι σε θέση η Επιτροπή, θα έχει την εξουσία, θα έχει την δύναμη να αντιταχθεί σε αυτέ τι πολιτικέ επιλογέ. Αυτό θα το κρίνετε εσείς που είστε οι Το ίδιο ισχύει για τις ε, κυρώσεις ή και για τους ελέγχους. Ή ισχύουν τα πάντα για όλους, τα ίδια για όλους, δηλαδή στρατηγικά σχέδια μέσα στα οποία ορίζουν τα κράτη-μέλη, τα συστήματα ελέγχων και τα ελάχιστα επίπεδα ελέγχων, τα επιβάλλει σε ένα ελάχιστο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό μπορεί να γίνει με μια κατεξουσιδότηση πράξη. Τότε γιατί όμω να μην το αποφασίσουν οι συνομοθέτε ω βασικό στοιχείο αυτό, πολύ βασικό και απαραίτητο, για την αξιοπιστία του συστήματος και για το σύστημα συμμόρφωσης που είπε και ο κύριος Μέγκελε ότι και νομίζω ότι σε αυτό απαντάμε λίγο και στις ε, προτάσεις ε, ή στις θέσεις του κύριου Ντόντα. Εάν λοιπόν έχουμε έναν οργανισμό πληρωμών, πιστοποίησης, εθνικό οργανισμό δηλαδή, με υπό την ευθύνη του την επαλήθευση, τον έλεγχο και την εξασφάλιση, χριστό, εξασφάλιση χρηστών δαπανών του δημόσιου χρήματος και θα μπορεί άρα αυτός ο οργανισμός να λέει ότι είναι ελάχιστο το ποστό του σφάλματος και, και παραμένει ελάχιστο και μηδαμινό, τότε γιατί να μην έχω ένα κοινοτικό σύστημα και να μπορώ να επαληθεύσω ότι και πάλι σε, ε, με χρηστό τρόπο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα δαπανώνται τα χρήματα της ΚΑΠ. Αποτελέσματα. Ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Τι είναι ως αποτελέσματα. Πόσα εκτάρια θα επαχθούν σε ένα συγκεκριμένο μέτρο ή θέλουμε κάτι παραπάνω, δηλαδή το μέτρο αυτό μέσα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο του κράτους μέλους κλπ. θα προσμετρά και τον αντίκτυπο για το περιβάλλον ή τη γενική οικονομία του κάθε μέτρου. Γιατί αν είναι μόνο στατιστική μέτρηση, αριθμητική μέτρηση, νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε να συζητούμε εδώ πέρα λέγοντας ότι έχουμε δύο-τρει εκτάρια που υπάγονται στο τάδε μέτρο, Χωρί όμω να είμαστε σε θέση να πούμε τι είδου αντίκτυπο έχουν φέρει για το περιβάλλον, για τον πολίτη, για την οικονομία. Όπου θα πούμε πάλι, μα η πολιτική αυτή δεν, δεν είναι πολιτική αποτελεσμάτων και θα μας πείτε εσείς, μα πάλι χάσαμε το στόχο μας. Όχι, οι δείκτες μέτρησης αποτελέσματος δεν προσφέρουν μετρήσιμα ή μετρούμενα αποτελέσματα. Ξέρω ότι έχει προχωρήσει αρκετά η δουλειά, αλλά μένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει και πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα. Και μια τελευταία παρατήρηση, για να απαντήσω στον κύριο Ντεκάστρο. Τα περιφερειακά οργανωμένα κρατή-μέλη, εθνικά σχέδια. Κοιτάξτε, δεν είμαστε Παπαδοπέδια, σε μια τέτοια περίπτωση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αναγνωρίσουν αυτήν, αυτό το χαρακτηριστικό της περιφερειακής οργάνωσης. Οπότε θα υπάρχει μια εθνική στρατηγική η οποία θα κατανέμεται σε διαφορετικές περιφερειακές στρατηγικές. Θα μου πείτε, έχει ενισχυμένο, ενέχει ενισχυμένο κίνδυνο για την προσέγγιση. Όντως, σε μητών. Αλλά τότε φτάνουμε, το αποτολμάμε να φτάσουμε μέχρι της εισαγωγή διαφορετικών περιφερειακών πολιτικών, κανόνων, κυρώσεων, ελέγχων κτλ. Δηλαδή όσα είναι τα, τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, καμιά κατοστή, θα έχουμε και σύνολα κανόνων, ελέγχων και κυρώσεων. Εγώ διατυπώνω το ερώτημα και πρέπει να δοθεί μια απάντηση σαφής για να ξέρουμε πού πάμε και σε θέση να διαχειριστούμε αυτή την εξέλιξη, αυτό το σύστημα. Και εάν κάτι τέτοιο θα είναι απλούστερο στη σχέση Επιτροπής και Κρατών Μελών μπορεί, γιατί την Επιτροπή να είναι πιο απλό. Για τον Γεωργό νομίζω ότι ή μη τι άλλο τα πράγματα δεν αλλάζουν, πάλι θα έχει κανόνες να τηρήσει. Ίσως οι κανόνε να είναι πιο στοχευμένοι σχέση με τις δικέ του ανάγκε. ανάγκες. Αλλά τότε α χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία. Να ξέρουμε τι αντιστοιχεί σε τι, ώστε όλοι να έχουν την ίδια βάση που θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν. Και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη θα έχουν και την καθαρή απόδοση και την πολυετή και την ετήσια αξιολόγηση. Πράγμα το οποίο το βλέπω αρκετά δύσκολο στη διαχείρισή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τσούμπακ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω σε ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Άγγλιο για παράδειγμα. Έκανε τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν τα εισοδήματα εκτός της γεωργικής δραστηριότητα, ορισμός του αγρότη και ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης. Άλλο ορισμός του αγρότη και άλλο ορισμός της ε, αγροτικής εκμετάλλευσης. Το πρόβλημα είναι ότι ένα τμήμα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνει και μη γεωργικά εισόδηματα, αλλά αυτό δεν ε, είναι το τέλος της ιστορίας. Πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ε, γίνονται απλώς για λόγους αναψυχής. Κάποιος αγοράζει μια αγροτική έκταση, περνάει εκεί το Σαββατοκύριακο και ασχολείται λίγο με τη γεωργία. Και από αυτή την άποψη είναι παραγωγή. Τοπική μεν, αλλά παραγωγή. Και αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται ψυχαγωγικά με τη Γεωργία. Επίσης, ε, τι γίνεται με τους συνταξιούχους Γεωργούς. Γιατί μπορεί ένα ε, γεωργό που βγαίνει στη σύνταξη να πουλήσει το μεγαλύτερο τμήμα τη αγροτική του εκμετάλλευση, αλλά ένα μικρό κομμάτι να το κρατήσει για να συνεχίσει παρόλα αυτά και τη συνταξιούχο την ε, γεωργική του δραστηριότητα. Και αυτέ οι εκμεταλλευσει είναι γεωργικέ εκμεταλλεύσει και το πιο ευαίσθητο θέμα είναι οι κερδοσκοπικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί στην περίπτωση Πολωνίας, για παράδειγμα, από 3.500 ζλότη ε, το 2004 είναι, έχει φτάσει στα 40.000 ζλότη ε, σήμερα. Οπότε υπάρχει μια κερδοσκοπία που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της τιμής των ε, αγροτικών γεών. Το θέμα είναι αυτοί που κερδοσκοπικά, για κερδοσκοπικούς λόγους αγοράζουν αγροτικές εκτάσεις, εμπίπτουν στον ορισμό του αγρότη. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αποκλειστούν από τον ορισμό του πραγματικού αγρότη, παρόλο που εμπίπτουν στον ορισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης, ε, βιολογική γεωργία. Και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πρακτικά. Η πλειοψηφία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των παραγωγών δεν ε, ταυτίζεται με τα οικολογικά αποτελέσματα της γεωργικής δραστηριότητας ή με άλλα περιβαλλοντικά μέτρα. Για τις φιλοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες, το βασικό κριτήριο που καθοδηγεί το Γεωργό είναι το οικονομικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα. Και κατά πόσο τα έσοδα, οι που λαμβάνει υπερισχύουν των δαπανών που θα κάνει για τα περιβαλλοντικά μέτρα. Το οικονομικό κριτήριο λοιπόν είναι αυτό που χρησιμοποιεί για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες ο αγρότης κατά κανόνα. Και μετά από πέντε χρόνια εφαρμογή ε, του συστήματο αυτού των περιβαλλοντικών μέτρων δεν έχουμε ε, μεγάλο ωφέλη στην Πολωνία. Εγώ είμαι επιστήμονας και από αυτή την άποψη έδωσα τις απαντήσεις μου και εντάξει μπορεί να γενικεύω μερικές φορές γιατί μπορεί όντως να υπάρχουν κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ε, εφαρμόζουν πιο, διασταλ, πιο συσταλτικά αυτό τον ε, ορισμό και πραγματικά δεν χρησιμοποιούν μόνο οικονομικά κριτήρια για τις περιβαλλοντικές ε, δραστηριότητες, αλλά οι περισσότερες νομίζω εκμεταλλεύσεις καθοδηγούνται από τέτοια κριτήρια. Επίσης, κάποιο άλλο στοιχείο που δεν αναφέρθηκε, η στέρηση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα. Γιατί μπορεί να γίνονται επενδύσεις, αλλά τα θετικά αποτελέσματα, τα οικονομικά των επενδύσεων φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση. Και αυτό επιβαρύνει τον Γιώργο που χρειάζεται να ζητήσει δάνειο. Αυτή η καθυστέρηση εμ, ενοχλεί πολύ τους Γιώργους. Και αν στόχος ε, της γεωργία είναι η παραγωγή ασφαλών τροφιμών, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργού και να τους απαλλάξουμε αυτά τα από, από τα αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης. Επίσης, ε, τα, μελ, τα με, η, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 άλλαξε τα δεδομένα και άλλαξε και τη θέση του παραγωγού. Οπότε θα πρέπει όλα τα κριτήρια που ανέφερε ο κύριος Αντριέ ε, να ισχύσουν και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή, ο γεωργός κατά την αγροτική του εκμετάλλευση να έχει μία προβλεψιμότητα στις δράσεις του, να γνωρίζει τι περιμένουν από αυτόν και να μπορέσει να προετοιμαστεί. Θέλει λοιπόν την προβλεψιμότητα που εξασφαλίζουμε και σε άλλους τομείς και θα πρέπει να ξέρει ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχει η παραγωγή του σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα κριτήρια του νέου μοντέλου υλοποίησης. Επίσης, στόχος των νέων μέτρων είναι ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διατυπώσεων. Η απλούστευση και η πιο γρήγορη λήψη των διοικητικών αποφάσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο απλοποίησης θα πρέπει να συντομευθούν, να συντομευθούν οι προθεσμίες για τη λήψη των αποφάσεων. Αυτό ενδιαφέρει πολύ τον ε, Γιώργο. Η απλούστευση, η πιο σύντομη εκαθάριση των λογαριασμών, όλα αυτά είναι θετικά στοιχεία απλούστευσης. Ένα άλλο στοιχείο απλούστευσης ε, είναι ε, οι αυξημένες διατυπώσεις που χρειάζεται να τηρήσει. Αυτό δεν έχει αλλάξει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να διορθωθεί, να μην αυξάνονται συνέχεια οι διοικητικές διατυπώσεις. Επίσης, ποιο είναι το κοινό στοιχείο της κοινή γεωρικής πολιτικής. Ο προλαλής σας μίλησε για τον πρώτο πυλώνα, που είναι ο πραγματικά κοινό πυλώνας. Ένα μεγάλο τμήμα του πρώτου πυλώνα είναι η άμεσες ενισχύσεις με διάφορες παραλλαγές. Ο στόχος όμως είναι κοινό, παρόλο που η διαφορά στις ενισχύσεις είναι μεγάλη. Και παρά τα διαφορετικά σενάρια υλοποίηση στις διάφορες χώρες, όντως το σημαντικότερο στοιχείο της ε, κοινή γεωρικής πολιτικής είναι ο πρώτος πυλώνας. Υπάρχουν κοινά στοιχεία και υπάρχουν και διαφορές στην κοινή γεωρική πολιτική. Πάντως, είναι δύσκολο να φανταστούμε σήμερα μία ενιαία γεωρική πολιτική όταν έχουμε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση των γεωρικών μοντέλων. Αλλά δεν θα, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτόν τον κατακαιρματισμό. Αρκεί τα κριτήρια και οι στόχοι της κοινή γεωρικής πολιτικής να είναι ενιαία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμόνε, και εσείς πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά και τα χρησιμοποιώ για να σας πω πολύ σύντομα ότι με όλα τα μειονεκτήματα μπορούμε να βρούμε στην ε, νέα ΚΑΠ, πάλι θεωρώ ότι θα απλουστευτεί η δουλειά για τον Γιώργο μας και αυτό το βλέπω σαν πλεονέκτημα. Ίσως περισσότερη επικουρικότητα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η τελική απάντηση, είναι η λύση τελικά. Ε, όλα τα άλλα Είμαι πεπισμένο πως αυτοί που λένε ότι το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να βάλουμε, τον Γεωργό σε μια πιο δύσκολη θέση, να τον πιέσουμε περισσότερο σχέση με τα όσα θα έχει να υλοποιήσει και τις απαιτήσει των κρατών μελών, περιφερειακή οργάνωση και προγραμματισμό τη ΠΑΚ, ε, θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τα απαιτούμενα αποτελέσματα. σχέση με τη νέα ΚΑΠ και για να απαντήσω στις ερωτήσεις και τον προβληματισμό σας, ίσως βρισκόμαστε δεδομένου ότι όπου να είναι φτάνουν και οι ευρωεκλογές, βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή και άρα θα πρέπει να γίνει και μια νέα αξιολόγηση ενδεχομένω. Νομίζω ότι μπορώ να δώσω απαντήσεις στους προβληματισμούς σας, αλλά θεωρώ πως η νέα ΚΑΠ ε, χρειάζεται να προσαρμοστεί στα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα, αλλά πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες, με ποσοτική μέτρηση. Και αυτή είναι και η τρόποι που αναζητούνται, πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να αξιολογήσει την ΚΑΠ και τις προτάσεις των κρατών μελών. Επομένως, εδώ θα μπορούσε η λύση να είναι μια πιο πυκνή διαβούλευση με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Αυτό δεν ξέρω ότι θα είναι δύσκολο να πληθεί το σχετικό δίκτυο. Δηλαδή, περιφερειακές αρχές, επιτροπή, κράτη-μέλη. Ε, η υπερβολική βέβαια επικουρικότητα και οι νέε προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνουν ότι απαιτείται ένα νέο πλαίσιο για την επικαιροποίηση και την επαλήθευση των ε, μέτρων. οι επιδόσεις θα είναι δύσκολο να, να αξιολογηθούν, να μετρηθούν με βάση τους ευρωπαϊκούς στόχους. Εδώ είναι τα όρια που βλέπω εγώ. Και βλέπω δυσκολίες, άλλωστε το διαπιστώνουν και τα μέλη της Επιτροπής. Και θεωρώ ότι θα χρειαστούν τα εξή Στόχοι σαφεί, ειδικοί, ποσοτικά μετρήσιμοι, μετρήσιμοι τα αποτελέσματα και την τήρησή τους, μέτρα συνδεδεμένα με τους στόχους, σύνολο στόχων, ε, ε, δικτών συγγνώμη, με συγκεκριμένα αποτελέσματα και αντίκτυπο μετρήσιμο. Όλα αυτά λοιπόν μέσα σε στρατηγικά σχέδια για την ΚΑΠ μπορούν να αποτελέσουν μια γνήσια προσθεμένη αξία και τα κράτη-μέλη μπορούν να αξιολογηθούν με βάση τις επιδόσεις. Αυτά είναι στοιχεία νομίζω και όπως βλέπετε Πρόεδρε δεν εξάδελσα και το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια στιγμή. Τι σημαίνει δίκτες επιπτώσεων και ε, πολύ προηγμένοι δείκτες επιπτώσεων και αποτελεσμάτων. Τι ακριβώς εννοείται, γιατί δεν κατάλαβα όταν μιλήσετε για προηγμένους δίκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. Τι θα πει αυτό. Να σας πω ότι εννοώ. Εννοώ ότι ο δίκτης πρέπει να αντιστοιχεί σε δύο ε, όρια. Εάν δεν είναι προηγμένος ο δείκτης, δεν θα έχει ποτέ την πιστοποίηση Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως ο δείκτης θα πρέπει να περιλαμβάνει και την δυνατότητα να καταγράφεται, να αξιολογείται με τρόπο αποτελεσματικό, άρα θα δίνει και περισσότερη αξιοπιστία σε αυτό που κάνουν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Δηλαδή θα επιτρέπει την ε, ε υλοποίηση του ρόλου τους, του ρόλου τους και περισσότερη, ε, α, περισσότερη αξιοπιστία και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ξέρουμε δηλαδή ότι μπορούμε με το μέτρο αυτό να επιτύχουμε καλύτερα από ότι με οποιοδήποτε άλλο μέτρο αυτό το οποίο επιδιώκεται. Και επί τη ευκαιρία, μια και μου το προσφέρατε πάλι το λόγο, θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμη η αξιολόγηση κάθε έτος, αλλά μόνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί μόνο έτσι μπορούν να καταγραφούν τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε τους εμπειρογνωμονές μας και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω από τη λέξη κοινή στην κοινή γεωργική πολιτική, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα στη συζήτηση. Και ακούστηκε το ποσοστό του 73% των ε, δαπανών ε, που ε, καταβάλλονται με κοινό τρόπο. Έχουμε διάφορα ιστορικά μοντέλα με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Έχουμε, για παράδειγμα, ενισχύσεις στην, στην Πολωνία. Και μάλιστα σε κάποια κράτη-μέλη καταβάλλονται περιφερειακά και έτσι έχουμε διαφορετικό σύστημα. Έχουμε κάποια κράτη-μέλη τα οποία ε, φτάνουν ε, το ε, συνολικό ποσοστό των συνδεδεμένων πληρωμών, άλλα κράτη-μέλη δεν έχουν καθόλου. Μερικά κράτη-μέλη εφαρμόζουν το κάπινγκ, αλλά όχι. Κάποια κράτη-μέλη ανέρχονται στο 30%, αλλά παραμένουν γύρω στο 6-7%. Και μάλιστα έχουμε ένα προαιρετικό στοιχείο όσον αφορά τους μόνιμους βοσκότοπους. Ε, αυτό ε, προκύπτει από τον κανονισμό Omnibus. Ακόμα δηλαδή και ο ορισμός των μόνιμων βοσκότοπων δεν είναι πια κοινό. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Και δεν το λέω αυτό για να σας δείξω ότι η πολιτική αυτή δεν αξίζει αντιθέτως. Αλλά δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να πιστέψουμε ότι έχουμε μια πολιτική η οποία είναι ίδια παντού. Και κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει και αλλιώ, διότι 27 κράτη-μέλη έχουμε, δεν ξέρω πόσες περιφέρειες έχουμε. Και η Σικελία διαφέρει πολύ από τη Φιλανδία. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφορές. Το ερώτημα είναι θα πρέπει ε, αυτή η ευελιξία να ισχύει διαπαντός ε, ή θα πρέπει η ευελιξία να βασίζεται σε αναλύσεις, αναλύσεις SWOT, αναλύσεις αναγκών, ε, διαλόγους με όλους τους ενδιαφερόμενους ε, και μια ε, προσεκτική διαδικασία από πλευρά της Κομισιόν. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μου παρέμβαση ότι με το νέο σύστημα το κάπα στην κοινή γεωργική πολιτική θα είναι πιο μεγάλο από ότι είναι σήμερα. Θα είναι δηλαδή πιο πολλά τα κοινά στοιχεία. Και πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, με ποια στοιχεία τα ανέφερα. Τρεις βασικούς στόχους, ε, εννέα επιμέρους ειδικού στόχους, ε, καθώς και ανάλυση SWOT και ανάλυση των ε, αναγκών καθώς και κάποιους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη, καθώς και ε, τα συστήματα διακυβέρνησης που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και κατόπιν θα έχουμε την διαδικασία έγκρισης που θα τα συνδυάζει όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σειρά βημάτων ε, που ε, πρέπει να κάνουμε κάθε φορά για την έγκριση του σχεδίου. Άλλωστε είναι προνόμιο του νομοθέτη να προσθέτει προϋποθέσεις ε, στον κατάλογο αυτών. Εάν θεωρείτε ότι δεν είναι κοινή, αρκετά κοινή γεωργική πολιτική, τότε ε, και αυτό θα αποτελέσει η τμήμα της όλης διαδικασίας. Κύριε Ντάντε, ρωτήσατε πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα εφαρμόζεται η κοινή γεωργική πολιτική με τον ίδιο τρόπο παντού. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ούτε σήμερα, ούτε στο μέλλον θα μπορούμε. Αν δείτε την ετήσια μας έκθεση θα διαποστήσετε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη με υψηλά ποσοστά λαθών και άλλα με πολύ χαμηλά ποσοστά. Παρά τις προσπάθειές μας ε, να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση στις περιπτώσεις των υψηλών ποσοστών λαθών. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, οι βασικές προϋποθέσεις στα διάφορα κράτη-μέλη διαφέρουν. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και αυτό δεν θα αλλάξει στο νέο σύστημα. Το νέο σύστημα όμως θα λειτουργεί με βάση άλλες παραμέτρους και την ομότητα και την κανονικότητα θα την αφαιρέσουμε από το επίπεδο του δικαιούχου, διότι πιστεύουμε ότι αν το διατηρήσουμε αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε τον φαύλο κύκλο όλο και πιο αναλυτικών κανόνων, πιο αυστηρών ε, ελέγχων και πιο αυστηρών κυρώσεων, διότι το κάθε επίπεδο διακυβέρνησης θα θέλει να φροντίσει ε, να είναι αδιάβλητο. Αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τις περιφέρειες δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλο, διότι ήδη έχουν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και έχουν μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό. Και μάλιστα ο Επίτροπος Χόγκαν συζητάει ακριβώς αυτό το θέμα με τον Ιταλό Υπουργό Γεωργίας και τις περιφέρειες και έχουμε παρόμοιες επαφές με άλλα αποκεντρωμένα ή ομοσπονδιακά κράτη-μέλη όπως είναι η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία και δεν πιστεύω ότι δεν μπορούν να λυθούν ε, τα θέματα αυτά που αφορούν τις περιφέρειες. Όσον αφορά το θέμα των επιδόσεων που αναφέρθηκε, προτού δώσω το λόγο στον συναδελφό μου, θα ήθελα να καταστήσω το εξής σαφές. Μιλάμε για δείκτες. Μιλάμε για δείκτες ε, που πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα του δείκτη ε, και την σκοπιμότητα χρήσης του. Υπάρχει δηλαδή ένα θέμα αποτελεσματικότητας και φυσικά υπάρχουν δείκτες επιδόσεων οι οποίοι μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στους σκοπούς των προτάσεων, ε, αλλά μπορεί να είναι τόσο επαχθείς που να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Στην πρόταση λοιπόν πιστεύουμε ότι έχουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στη σκοπιμότητα του δίχτυα από τη μία μεριά και την ε, σκοπιμότητα όσον αφορά τις δαπάνες από την άλλη μεριά. Ο συνάδελφός μου όμως θα ήθελε να προσθέσει κάποια πράγματα. Πέντε λεπτά μόνο, όχι παραπάνω. Σας ευχαριστώ και ακόμα λιγότερο όσον αφορά το σημείο αυτό. Η επιλογή δίκτυ. Όταν ακούω ότι... Ε, όταν ακούω αυτά που λέτε σχετικά με τον ε, αντίκτυπο, εν μέρη μπορώ να συμφωνήσω μόνο, διότι το σύστημα αυτό προβλέπει πρόοδο ε, όσον αφορά την επίτευξη ενός στόχου και από την άλλη έχουμε τον αντίκτυπο. Ο δείκτης αντικτύπου υπολογίζει το τελικό αποτέλεσμα επιτόπου στην πράξη. Δηλαδή, αν ένα κράτος μέλος πιστεύει ότι για να φτάσει το στόχο του υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες ε, όσον αφορά τον, τον οργανικό άνθρακα, μπορεί να, ε, του εδάφους, ε, μπορεί να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα και αυτό θα φαίνεται ε, στο output, στο ποσοστό των ε, διαφόρων φορέων. 2-3% ε, του εδάφους ε, μπορεί να καλύπτεται από αυτή την υποχρέωση και τελικά η προσπάθεια αυτή θα φαίνεται και στον δίκτυ αντικτύπου. Όταν δηλαδή πάνε οι στατιστικοί να υπολογίσουν τον οργανικό άνθρακα στο έδαφος. Για να αποδείξει κανείς το πόσο γόνιμο είναι το έδαφος, δεν μπορεί να το κάνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία μακρόχρονη Πρέπει όμως κάποια στιγμή να ξεκινήσει. Νομίζω λοιπόν ότι η πολιτική όσον αφορά τον αντίκτυπο είναι σαφής και είναι και φιλόδοξη. Όσον αφορά την ε, εσωτερική σύγκληση πληρωμών ε, ανάμεσα στους γεωργούς, αυτό είναι αποτέλεσμα συναπόφασης κατά την τελευταία μεταρρύθμιση θα ήθελα να αναφερθώ στον δικτυ i I24 με τον τίτλο Δικαιοσύνη. Το συζητάμε αυτό αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες σε σχετικά με το τι σημαίνει ο κάθε δείκτης, πώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται, ποια θα πρέπει να είναι η μεθοδολογία. Ο δείκτης αυτός μπορεί να δείχνει το ποσοστό γεωργών που λαμβάνουν τη στήριξη σύμφωνα με τον κανόνα 80-20, 80%-20%. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά αυτή τη στιγμή με τα κράτη-μέλη για τους δείκτες, διότι είναι οι πρώτοι που θα καταρτήσουν σχεδρικό σχέδιο. Θα κοιτάξουν τα νούμερα και θα, θα εκπονήσουν τελικά μια έκθεση. Καταβάλουν λοιπόν πάρα πολύ χρόνο τα κράτη-μέλη, καταβάλουμε εμεί πολύ χρόνο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε όλε τι λεπτομέρειε. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έρθουμε εδώ να σα εξηγήσουμε πού βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτή. Διότι νομίζω ότι αν υπάρχει περισσότερη σαφήνεια, καλύτερη κατανόηση, τότε ε, θα ε, διασκεδαστούν πολλοί από τους φόβους που ακούω σήμερα. Ευχαριστώ ο κύριος και μίλησε για την κερδοσκοπική αγορά γεών. Ε, το θέμα αυτό συζητήθηκε εκτενώς και είχαμε και μία ειδική έκθεση νεαρών επιστημόνων από την Ολλανδία και έχουμε και την έκθεση της κυρίας Νόιχλ. Οπότε δεν είναι ένα θέμα που πέρασε παρατήρητο το θέμα της κερδοσκοπικής αγοράς γεωργικών εκτάσεων. Ε, επίσης, έχουμε έχουν προετοιμαστεί, έχουν ήδη εκπαιδευτεί πολλά ε, σχέδια και στον πρώτο πυλώνα και εκεί υπήρχε διαφοροποίηση. Οπότε υπάρχει και ένα κενό στοιχείο, αλλά υπάρχουν πολλές διαφοροποίησεις. Τώρα, το, η διαφύλαξη αυτού του κοινού στοιχείου περνά από τις ε, από τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την αξιολόγηση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αναλάβει μόνη της όλα και να μονοπολίσει τις δραστηριότητες, ούτε να περιορίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στα θέματα αυτά. Γιατί σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, αλλά δεν θα πρέπει να παραγωνίσει τους νομοθέτες, ε, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Δεν θα πρέπει όμως να μένει στο περιθώριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το ίδιο ισχύει και για την φάση της εφαρμογής. θα πρέπει στην εφαρμογή και στις αξιολογήσεις που θα γίνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παραμεριστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί και η Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσουν τη γνώμη τους για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι προσυζήτηση. Χρειάζεται διάλογος, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε επαρκή διάλογο. Ούτε για την παραγωγή των τροφίμων, ούτε για το διάλογο μεταξύ των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας. Κύριε Φλάναγκαρ, παρακαλώ ένα λεπτό μόνο. Θα ήθελα να ε, μιλήσω για ένα θέμα στα διάφορα όταν φτάσουμε εκεί, αν έχουμε φτάσει εκεί. Προτού κινητοποιηθεί το άρθρο 50, μας είπαν στην Επιτροπή τούτη ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε το Brexit μέχρι να ενεργοποιηθεί. Δεν θα μπορούσαμε να συγκαλέσουμε ειδική επιτροπή για να συζητήσουμε τις ε, συνέπειες. Σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, η Ιρλανδία και οι 16 κομιτείες ε, ε, της βόρειας πλευράς του νησιού θα ε, αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές συνέπειες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω στην Κομισιόν πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω. Θα συζητηθεί το θέμα αυτό την Πέμπτη ή θα ζητηθεί σε μελλοντική συνεδρίαση της Άγκρη διότι δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο για τη χώρα μου αυτή τη στιγμή από αυτή την απειλή, από την κατάσταση που μας απειλεί σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνίας η κυβέρνησή μας μας λέει λίγα πράγματα για το τι μπορεί να κάνει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως ε, ε αρμόδια επιτροπή στο Κοινοβούλιο αυτό για το θέμα αυτό, μπορεί η Κομισιόν να μας πει τι θα κάνει σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, διότι ε, γνωρίζουμε ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα χάος στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Η επόμενη μας συνεδρία θα γίνει στις 7 Μαρτίου, δηλαδή πολύ σύντομα. Στις 18 όμως Μαρτίου, στη μεθεπόμενη μας συνάντηση, θα έχουμε περισσότερες ε, ε, ίσως πληροφορίες για τα θέματα αυτά του Brexit από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα έλεγα αυτά τα θέματα να τα αφήσουμε και τις 18 Μαρτίου για τη μεθεπόμενη συνεδρίαση, γιατί ε, κάποιες αποφάσεις θα ληφθούν όχι σε δικό μας επίπεδο, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και εμείς αυτά τα θέματα. Για να περιορίσουμε αυτή την ανησυχία που επικρατεί. Ελπίζω να ληφθούν ε, αποφάσεις σωστές για τα θέματα αυτά. 7 Μαρτίου η επόμενη μας συνεδρίαση, 9 με 12.30 και η μεθεπόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 18 Μαρτίου. Ε, χαίρομαι που είχαμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Σπάνια έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου και ε, δεν αναγκάζομαι να κόβω το μικρόφωνο ή να περιορίζω το χρόνο γόρευση πυρογνωμόνων ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Ευρωβουλευτών. Χαίρομαι που σήμερα είχαμε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου. Σας ευχαριστώ και κηρύσω το πέρα τη συνεδρίασή μας. Καλώς βράδυ.